Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, γιατί είναι 3 και 5 και η ημερήσια διάταξη είναι βεβαρημένη σήμερα το απόγευμα, διότι έχουμε ανταλλαγή απόψεων, το σημείο 24, με την κυρία Αλτζιμάντα Παμπετίνσκινιε, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Λιθουανική Λιθουανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητή κυρία Υπουργέ, σας δίνω το λόγο για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη. Ξέρω ότι έχετε ήδη συναντηθεί με διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής μας όταν μετέβησαν στη Λιθουανία για επίσκεψη, είχατε διμερείς επαφές και χαίρομαι διότι σας βλέπουμε ξανά επισήμως στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να κάνω μια ανασκόπηση των βασικών προτεραιοτήτων της Λιθουανίας στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Βεβαίως, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σήμερα, αφού το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί ε, τα συμφέροντα 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα επιδιώξουμε ε, μια συνεργασία επικοδομητική, παραγωγική και αμοιβαίως ε, ωφέλιμη. Είναι η πρώτη φορά που η Λιθουανία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό είναι εξαιρετική πρόκληση για τη χώρα μας, αλλά και εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε την χώρα μας στην Ευρώπη. Τους έξι επόμενους μήνες η προσοχή μας θα στραφεί γύρω από τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα κράτη-μέλη με σκοπό να πετύχει η Προεδρία μας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Λουθουανία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει μια ομαλή και συνεχή νομοθετική διαδικασία. Θα είναι ένας δίκαιος και αμερόληπτος ε, διαμεσολαβητής ο οποίος θα προσπαθήσει να εμπλέξει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα επιδιώξουμε τους στόχους ε, της, ε, των τριών προεδριών, της προηγούμενης από εμά και της δικής μας και της επόμενης από εμά, Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα. Και θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο σημαντικά καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να γίνουν οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών της ακόμα πιο ε, δεσμευτικές και να ξεπεράσουμε τις οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, θα ενισχύσουν την απασχόληση, θα βελτιώσουν την ενιαία αγορά, θα διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα ενισχύσουν την οικονομική και νομισματική ένωση. Μια ένωση η οποία κατά την άποψή μας πρέπει να είναι στεναρή όχι μόνο από οικονομική, σκοπιά, από οικονομική σκοπιά αλλά και από κοινωνική σκοπιά. Έχοντας αξιολογήσει την κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχοντας ε, ξεπεράσει με επιτυχία την ε, οικονομική κρίση που είχε διανύσει, που είχε αντιμετωπίσει, η, Λιθουανία, η Λιθουανία θα δώσει έμφαση στη δημιουργία μιας αξιόπιστης, αναπτυσσόμενης και ανοιχτής Ευρώπη, Ευρώπης. Επιθυμούμε ως Προεδρία να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, να διασφαλίσουμε επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση και να εδραιώσουμε πραγματική ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ως προς τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ σε καλύτερες ε, ευκαιρίες απασχόλησης, ε, κυρίως για τους νέους. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτησή της απόφασης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Πολύ συχνά, λόγω έλλειψης εργασιακής εμπειρίας και λόγω απουσίας επαρκών προσόντων ε, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι νέοι ε, έχουν πολύ περισσότερα εμπόδια να ξεπεράσουν ε, κατά την αναζήτηση εργασίας. Και μάλιστα η οικονομική κρίση γίνεται κοινωνική κρίση. Οι κοινωνικώς ευπαθείς νέοι αποκλείονται όλο και περισσότερο και τίθενται στο περιθώριο. 8 εκατομμύρια τώρα είναι οι νέοι που δεν βρίσκονται ούτε σε απασχόληση, ούτε σε κατάρτιση, ούτε ε, ε, σε σπουδές. Ε, είναι ένας αριθμός ο οποίος έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό η, όλο, τα όλο και μεγαλύτερα χρονικά διαλύματα μεταξύ εκπαίδευσης και έναρξης εργασίας, η πολύ συχνή απασχόληση, ε, η και οι μεγάλες περίοδοι χωρίς δουλειά θα έχουν αντίκτυπο αρνητικό μακροπρόθεσμο στις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και στο επίπεδο της αμοιβή που θα πετύχουν οι νέοι. Όλα αυτά ε, μπορεί να οδηγήσουν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Άλλες αρνητικές συνέπειες είναι η απομόνωση, η κοινωνική απομόνωση, η εμπλοκή σε επικίνδυνες ή ακόμα και ποινικώ αξιόπινες δραστηριότητες, η μη ασταθής ε, υγεία σε ψυχολογικό αλλά και οργανικό επίπεδο και η αποξένωση από τη δημοκρατική διαδικασία μεταξύ άλλων. Επομένως, ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα εστιάσουμε την ε, προσπάθειά μας στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων. Θέλουμε να προετοιμάσουμε ετοιμαστούμε καταλήλως για το σύστημα εγγυήσεων ε, προς τους νέους, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2014 και το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα οργανώσουμε συζητήσεις με τους υπουργούς και με τους κοινωνικούς εταίρους για να μοιραστούμε βέλτιστες ε, πρακτικές και να αναλάβουμε κοινέ δράσεις επί Βεβαίως οι, το, οι υπηρεσίες έβρεσης εργασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες έβρεσης εργασίας αλλά και ε, απασχόλησης των κρατών μελών θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Οφείλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, για την πρόταση, την πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις περιόδους μαθητείας ε, που θα βασίζονται αυτή, αυτές οι περίοδοι μαθητείας στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας, η οποία υπογράφει την οποία υπέγραψαν οι αρμόδιες αρχές ως κείμενο στις αρχές αυτού του μήνα. η Λιθουανία θα προσπαθήσει να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των νέων και κυρίως των νέων που δεν, ε, δεν σπουδάζουν, δεν έχουν βρει δουλειά και δεν ακολουθούν προγράμματα κατάρτισης. Ε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eurofound, λόγω της μη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει 150 δις ευρώ κάθε χρόνο από πλευράς κοινωνικών εισφορών που δεν καταβάλλονται και φόρων που δεν εισπράττονται ε, από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται προφανώς. Επομένως, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Νέων θα ε, ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα του αποκλεισμού των νέων και επιδιώξουμε να υιοθετηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα αναλύουν ε, τις αρχές που προτείνονται στα κράτη-μέλη και θα ασχοληθούμε και τα μέσα για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης όλων αυτών των νέων. Ε, κλείνω αυτό το θέμα των καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης ε, αναφερόμενη στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σκοπός ε, της πρότασης αυτής ήταν η βελτίωση, ήταν οι περισσότερες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και καλών πρακτικών ώστε να ταυτοποιείται, να εντοπίζεται καλύτερα η αδήλωτη εργασία και να υπάρξουν μέτρα ε, λειτουργικά, επιχειρησιακά. Είναι πολύ σημαντική ε, πρόταση και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει συνένεση στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να χαιρετήσω το προηγούμενο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ διότι ε, δούλεψε εντατικά για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων και υιοθέτησε κοινή θέση ε, ως προς το τόσο σημαντικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, γιατί διείστανται αρκετά οι απόψεις των κρατών μελών. Ε, όμως είναι ένα θέμα επίγον και είμαστε αποφασισμένοι να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί, να λειτουργήσει ε, το Ταμείο αυτό από τις αρχές του 2014. Στα τέλη Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη βελτίωση της ομοιόμορφης εφαρμογής και υλοποίησης και σεβασμού τήρησης, αν θέλετε, του θεμελιωδός δικαιώματος της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις ε, σε βάρος ε, των εργαζομένων στα κράτη-μέλη επί τη βάση της υπηκότητάς τους. Ωστόσο, στην πράξη, οι μετανάστες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν άμεσες διακρίσεις αλλά και έμεσες διακρίσεις λόγω της ηθαγενειάς τους. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε ε, την ε, δουλειά που έχει ε, ξεκινήσει με την οδηγία που έχει ξεκινήσει για την οδηγία των εργαζομένων με απόσπαση ώστε να βελτιώσουμε την παροχή των υπηρεσιών, να προστατεύσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους και να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα επιδιώξουμε συμφωνία με το Συμβούλιο και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το ε, Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που έχουν ε, ξεκινήσει οι Ιρλανδοί συνάδελφοι ως προς την εναρμόνιση των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Περιμένουμε και τα δύο θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν επικοδομητική προσέγγιση ε, για όλα αυτά τα θέματα ε, της υγείας της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και θα έχουμε τις απαραίτητες ε, τροποποιήσεις που χρειάζονται για την ταξινόμηση, την σήμανση, την ετοκετοθεσία, τη συσκευασία των χημικών. Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική συνεργασία γιατί τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα από την τεχνική πλευρά και πρέπει να αναλύσουμε όλες τις δυνατότητες προσεκτικά. Ε, προτιθέμεθα επίσης να ξεκινήσουμε συζήτηση για μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαγραφή των εξαιρέσεων των ναυτικών. Ε, εξαιρέσεις που υπάρχουν σε ορισμένες οδηγίες που έχουν να κάνουν με το εργατικό δίκαιο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση όλων των ε, πολιτικών. Έχουμε το SIP, ε, το Social Investment Package θα τονίσουμε τα συμπεράσματα του πρόσφατου, του τελευταίου ε, Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, το οποίο ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν εφαρμοστικές δράσεις προκειμένου να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο ε, το πακέτο αυτό των κοινωνικών επενδύσεων. Στις 11 και 12 Ιουλίου θα συζητήσουν οι Υπουργοί στο άτυπο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ με θέμα κυρίως την ε, εφαρμογή των συστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο. Πολύ μεγάλο ρόλο στην ε, ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης διαδραματίζει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους πιο ενδεείς. Παρόλο που η Ιρλανδική Προεδρία δεν κατάφερε να πετύχει τελική ε, συμφωνία για το Ταμείο αυτό, η πρόοδος που σημείωσε η Ιρλανδική Προεδρία είναι σαφέστατα απτή και πάρα πολλά σχόλια έκαναν τα κράτη-μέλη και λήφθησαν υπόψη από την Ιρλανδική Προεδρία. Αυτό το οποίο εκκρεμεί λοιπόν είναι να ε, συμφωνήσουμε στο κατά πόσο η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ταμείου θα είναι υποχρεωτική ή θα είναι σε θελούσια βάση. Και μένει να συμφωνήσουμε και για το μέγεθος του Ταμείου. Οι συζητήσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με τα κοινωνικά ζητήματα δείχνει ότι διαγράφεται ε, σαφέστατα μία ομάδα χωρών αρκετά σημαντική η οποία θεωρεί ότι η επανεργοποίηση των μέτρων που στοχεύουν να ετοιμάσουν τους ανθρώπους καλύτερα, να τους προετοιμάσουν για την αγορά εργασίας, είναι και ο καλύτερος τρόπος για την εξάλληψη της φτώχειας ε, στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ε, σύμφωνα με αυτή την ομάδα των κρατών μελών, τα μέτρα από που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι και τα πιο ε, κατάλληλα για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό. Ε, ε, μια άλλη ομάδα κρατών μελών εγκρίνει την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των κρατών μελών στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας ή Αρρωγής και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας αλλά μόνο στο πλαίσιο της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητο αυτό το μέτρο για τη μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη και το ίδιο πιστεύουν αρκετοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ποια είναι τα καλύτερα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας οι διαφορές στην κοινωνική πολιτική του κάθε κράτους μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές. Η Λιθουανία έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία που έχει αυτό το Ταμείο για τους πολίτες των κρατών μελών. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση αποδεκτή. Αποδεκτή ε, από όλα τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα από τα μελήματα που, που έχουμε και θα τα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα χωρίς ε, να χρονοτριβήσουμε. Ε, έρχομαι τώρα στις συντάξεις και έχουμε ε, την οδηγία για την κτήση και την διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Είναι ένα έγγραφο του 2005 και τελικά τα κρατημέλη επιτέλους έχουν φτάσει σε μια κοινή θέση. Η Ιρλανδία έκανε εξαιρετική δουλειά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στον τομέα αυτό και πέτυχε έναν αποδεκτό ε, συμβιβασμό. Οι αρχικές διαφωνίες για τη νομική βάση της ε, οδηγίας, για τον χρόνο αναμονής μέχρι ότου γίνεται κανείς μέλος αυτού του συνταξιδοτικού προγράμματος, αλλά και για την περίοδο κτήσης, απόκτησης των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων, ήταν πολύ ακαθόδη ζητήματα, τα οποία όμως επιλύθηκαν με συνένεση. Περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει συμφωνία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτή η τόσο σημαντική νομοθετική πράξη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Προσπαθώντας λοιπόν να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, περιμένουμε με ανυπομονησία τον οδικό χάρτη, το έγγραφο αυτό το οποίο ε, θα περιλάβει, θα περιλαμβάνει και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις μας. Ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό και θα εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή είναι δύο διαδικασίες που είναι αλληλοσυμπληρωματικές. Η μία ενισχύει την άλλη. Ε, δεν ε, συμβαίνει, δεν ισχύει η, το ότι η μία αποκλείει την άλλη η αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η όξυνση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι αυτό το οποίο τελικά και σε βάθος χρόνου σίγουρα απειλεί την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γι' αυτό και πρέπει να βρεθεί ένα σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών μέτρων και των κοινωνικών στόχων. Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πρακτικής διαχείρισης, ώστε να είναι αυτή πιο χρηστή, έχουν ήδη γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην κοινωνική σφαίρα πλέον. Και σε ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. τη διάρκεια της προεδρίας μας θα επικεντρωθούμε στο στόχο των ίσων δικαιωμάτων και τις προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση του στόχου αυτού. αποτελεσματική διακυβέρνηση και υλοποίηση των κανόνων απαραίτητη προκειμένου να επιληθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα ανδρών και γυναικών σαν εγκάρση αποτεραιότητα σε όλους του τομεί πολιτικής, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Έχουμε σε εκ τούτου επιλέξει ε, για τον κρίσιμο χώρο των ε, θεσμικών μηχανισμών της πλατφόρμας του Πεκίνου για δράση, και αποτελεσματική των θεσμικών μηχανισμών είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότητα ώστε αυτή να καταστεί πραγματικότητα και όχι μόνο ε, γράμμα στον νόμο. το σύμφωνο, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Δύο Φύλων και η Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνουν αρχέ καλή διακυβέρνηση ω απαραίτητη προπόθεση για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων για την ισότητα των φύλων που έχουν διατυπωθεί σε αυτά τα έγγραφα. Όπως ε, έχουμε επιλέξει εμείς ως Προεδρία, θα καταστήσουμε ε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση σε επίπεδο Συμβουλίου συμπερασμάτων για τους θεσμικούς μηχανισμούς στην ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου Απασχόληση και Κοινωνικών Θεμάτων του Δεκεμβρίου. Επιπλέον δε, αποστηρίζουμε την επιδίωξη τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή για τη βελτίωση τη εκπροσώπηση των γυναικών στον χώρο τη λήψη αποφάσεων και συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, ε, προσπάθειε που έχουν ξεκινήσει άλλωστε και από την Ισλανδική Προεδρία. Στο χώρο τη ισότιμη ε, μεταχείρισης συνεχίζουμε τι συζητήσεις για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία κατά των διακρίσεων, θα διακριτήσουμε ε, ευρύτερη συνενέση επίπεδο Συμβουλίου και επίση,. Θα επεξεργαστούμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένοντας βέβαια ε, ε, ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 26 Ιουνίου, με ιδιαίτερη με ιδιαίτερο μέλημα τη βελτίωση των μέτρων για την ενσωμάτωση του πληθυσμού των Ρωμά, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πολύ περισσότερο από ό,τι ποτέ. Έχουμε 6 εκατομμύρια Ρωμά που ζουν στην Ευρώπη. Και άρα είναι σημαντική ενσωμάτωση της κοινωνία όσο ποτέ. Έτσι λοιπόν, στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων ε, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ρωμάν στα κράτη-μέλη. Ξέρετε κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε για το εξάμεινο αυτό. Ένα εξάμεινο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη Λιθουανία. Κυρία Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά τώρα θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. ουσεμπρέστος τεξλός. Και ελπίζω θα μας στηρίξει στην επιτεύξη των στόχων μας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος με εντυπωσιάζουν τα επιτεύγματα που έχει μπροστά τη η Λιθουανική Προεδρία. Ελπίζω να μην εντυπωσιαστείτε κι εσείς από τον αριθμό των ερωτήσεων που θα σας υποβάλουν οι συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρώτα, με τον κύριο Ερή. Και μετά στου οριστές δημοκράτες, κύριε Πινκεβιτσούτε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό. Ήρθαμε μια κάποια καθυστέρηση. Ε, αλλά έχουμε ήδη την ευκαιρία να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο, γνωριζόμαστε. Έχω δει και παρακολουθήσει και τις πληροφορίες που έχουν ήδη ε, καταστεί γνωστέ σε σχέση με το πρόγραμμα τη Προεδρίας και χωρίς να θέλω να μακρηγορώ θα μου επιτρέψετε να εντυπώσω κάποιες ερωτήσεις για πιο συγκεκριμένα θέματα. Δύο υποθέσεις που έχει ε, κληρονομήσει από την προηγούμενη Προεδρία η Λιθουανική, το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων καταρχάς και Δεύτερον, η επιστημική βοήθεια για εκείνους που έχουν προσθέτει ανάγκη. Κατεπήγοντα ζητήματα, διότι πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα από τον Ιανουάριο. Έτσι λοιπόν μου φαίνεται κάπως ε, εξοραϊσμός της κατάστασης το να λέτε ότι υφίσταται απόκληση απόψεων. Υπάρχει μια ανασχετική μειονότητα αυτή τη στιγμή η οποία παρεμποδίζει την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Έχουμε εγκρίνει μια ε, αντιπροσωπεία διαπραγμάτευσης. Έχει σαφή εντολή για διαπραγμάτευση. Περιμένουμε να προχωρήσει μια κοινή θέση με στο Συμβούλιο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Έχετε λοιπόν κάποια ιδέα για το πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που λειτουργεί για την αντιμετώπιση των αμέσων κινδύνων, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει μια κοινή θέση στο Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Νέο στοιχείο επίσης είναι η καταπολέμηση της ε, παράνομης απασχόλησης και βέβαια ε, η ιδέα αυτή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, την υποστηρίζουμε. Θα πρέπει ωστόσο να δούμε βεβαίως και οι επιχειρηματίες πώς βλέπουν τις ε, προτάσεις. Θα τα συζητούμε όλα στο κοινοβούλιο για την ε, δυνατότητα μεταφοράς των σταξιδοτικών δικαιωμάτων. Έχουμε μια αντιπροσωπεία διαπραγματευτική εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια κοινή προσέγγιση, διατυπώσει ήδη και σας καλούμε να καταλήξετε το δυνατό σε μια συμφωνία. Και εν τέλει για το τομείο για την Παγκοσμιοποίηση. Με χαρά ακούμε τόσα είχατε να πείτε βεβαίως, αλλά ε, όλο μας λένε ότι δεν αρκούν τα χρήματα όταν ε, συζητούμε για προϋπολογισμό. Λοιπόν, ε, η, η ζήτηση αυξάνεται. Τα όσα αποφασίστηκαν είναι βέβαιο ότι δεν θα αρκούν ε, για τη χρηματοδότηση των αναγκών. Ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην αναλύεται όλο το πρόγραμμα της Λουφανικής ε, Προεδρίας έκαστος. Δεν θα τα καταφέρουμε διαφορετικά. Κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. E, Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και παρουσιάσατε με τόσο συνολικό και πλήρη τρόπο τις προτεραιότητές σας για να ολοκληρώσετε μια σειρά δραστηριοτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι οι λιθουανικές αρχές και οι υπάλληλοι δούλευαν για το σκοπό αυτό το συντομότερο δυνατό και ελπίζω να πετύχετε καλά αποτελέσματα. Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές σας, αναφερθήκατε αρκετές φορές στο ότι πρέπει να θυμόμαστε πως η κοινωνική διάσταση είναι αναγκαία στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, ακριβώς όπως και η ευημερία των πολιτών και ότι όλοι το χρειάζονται αυτό. Θέλω να θέσω καμιά σειρά ερωτημάτων που θεωρώ σημαντικές. Πρώτον, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. η απορρόφηση των πόρων και το ίδιο το Ταμείο έδειξε ότι χρειάζεται ότι χρειάζεται το Ταμείο αυτό για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόκειται για ένα ουσιαστικού χαρακτήρα μέτρο. Τι άποψη έχετε εσείς ως Υπουργός και το Υπουργείο σας σε ό,τι αφορά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο. Συζητήσαμε σήμερα το πρωί ότι πιστεύουμε πως τουλάχιστον το 25% του ταμείου, των Ταμείων Συνοχής πρέπει να πηγαίνει στο Κοινωνικό Ταμείο. Η Επιτροπή ωστόσο έχει διαφορετική άποψη και κράτη-μέλη έχουν επίσης διαφορετικές απόψεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνεισφορά της Λιθουανίας στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πετύχουν το 25%. Δεύτερον, είπατε ότι η προτεραιότητά σας είναι η μείωση της ενεργείας των νέων. Αναφέραμε το θέμα αυτό πολλές φορές. Αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής. Πέραν του περιορισμού της ανεργίας μεταξύ των νέων υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες. ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι. Αν μιλούμε για επιμήκυνση της ηλικίας συνταξιοδότησης, αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους. Εσείς ως Προεδρία τι θα κάνετε, κάτι ακόμα. Είπατε ότι το θέμα του mainstreaming ε, είναι πολύ σημαντικό στον τομέα αρμοδιότητά σας. Επίσης, μιλήσατε, μιλήσαμε χτες για ποσοστώσεις παρουσίας γυναικών σε μη εκτελεστικές διευθυντικές θέσεις. Πρέπει να σας πω ότι την οδηγία αυτή δεν υποστηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Θα σας ευχόμουν να επιτευχθεί κοινή συμφωνία μεταξύ κρατών μελών, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή του Κοινοβουλίου ακούγεται. Αλλιώ, εμείς δεν έχουμε, δεν έχουμε δυνατότητες να παρέμβουμε. Καλή επιτυχία σε εσά και σε όλους μας εδώ, γιατί θα το χρειαστούμε. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω ότι για το 25% Σήμερα η Κομισιόν είπε σαφώς ότι υποστηρίζει το αίτημα της Επιτροπής μας να ξανανοίξει ο φάκελος και να διατηρηθεί η αρχική πρόταση του 25%. Το Συμβούλιο είναι μόνο κατά. Μαριάν Άρκιν και μετά η Ντανούτα αγιά. Δεν σας περιέρισα το χρόνο, θα το κάνω και στην κυρία Άρκιν, αλλά μετά θα περικόψω. Εγώ θα είμαι σύντομη, πρόεδρε. Να καλωσορίσω την Υπουργό Καταρχά. ευχαριστούμε που ήρθατε και αφιερώνετε χρόνο σε εμά. Εκτιμούμε ε, την δουλειά σας. Σας είδα και στο Στρασβούργο βέβαια. Τέσσερις ερωτήσεις. Εγγύηση, ευρωπαϊκή εγγύηση νέων. το, το, το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει μια, ήδη μπήκε η παρέκκληση λόγω κρίσης που είναι μια μεγάλη αλλαγή πορείας. Η ερώτηση που σας θέτω, τι ήταν αυτό που επέτρεψε στην παρεμποδίζουσα μειοψηφία να μπλοκάρει τις συζητήσεις. Ανεργία νέων τώρα, έλειπα όταν παρουσιάστηκε τη θέση αυτή εμείς ε, από τη μεριά της ε, προσφοράς κάναμε πολλά. Από την πλευρά της ζήτησης εσείς έχετε να προτείνετε κάτι. Είπατε επίσης στην παρέμβασή σου κάτι πρέπει να γίνει στον κοινωνικό τομέα. Τι εννοείτε. Και τέλος γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια. Μίλησε η συνάδελφος, το ψηφίσαμε και σήμερα. Θέλω να ρωτήσω, η θέση στο Συμβούλιο ποια είναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδο στο ντοσχέ αυτό. Άλλοι δύο μιλητές και μετά κύριε Υπουργέ θα σας ε, δώσω το λόγο να απαντήσετε σε αυτή την πρώτη ομάδα ερωτήσεων που είναι ήδη μεγάλη. Ήταν το Ιγιοζιεύσκα και μετά ο Αλεχάντρος Σέρκας και μετά η Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον τόσο μας είπατε. Ελπίζω ότι θα έχουμε αρκετό, αρκετά επικοδομητικό πνεύμα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απόσπαση των εργαζομένων. Όπω ξέρετε, οι διαπραγματεύσει ε, στην Επιτροπή μα ε, έχουν κρατήσει αρκετό καιρό και παρά μια επικοδομητική προσέγγιση των πολιτικών ομάδων δεν ήταν φιερεί ε, σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Άλλωστε, ξέρω ότι και στο Συμβούλιο είναι αντίστοιχη αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα να ρωτήσω τη δική σα θέση και την κατάσταση, πώ βλέπετε τα πράγματα. Μια θετική προσέγγιση λοιπόν στην οδηγία αυτή. Και επίσης, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις κοινωνικές επενδύσεις. Με χαρά ακούω ότι η Επιτροπή μας ξεκίνησε τη δουλειά στα θέματα αυτά. Πολλές φορές υπογραμμίζουμε ότι οι κοινωνικές επενδύσεις είναι οργανωμένες, εφαρμόζονται μακροπρόθεσμα και μερικές φορές κάποιοι θεωρούν μόνο δαπάνες και όχι επενδύσεις. Αυτό, σε αυτό θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Κύριε Σέρκας. Καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ μας υποδεχθήκατε με πολύ θερμό τρόπο στο Βίλνιους. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το πρόγραμμα της Προεδρίας σας ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις συζητήσεις μας τότε. Θα ήθελα δύο αιτήματα να σας υποβάλω. Πρώτον, ο κύριος Φαν Ρομπόη υποσχέθηκε το Δεκέμβριο ότι τον Ιούνιο θα είχαμε ένα πακέτο για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με κοινωνικό πυλώνα. Πέρασε ο Ιούνιος και δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Πολύ φοβούμαι ότι ούτε το Δεκέμβριο θα υπάρξει κοινωνικός πυλώνας στην ΟΝΕ, εκτός και αν συνεργαστούμε με το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ και απαιτήσουμε να υπάρξει τέτοιος πυλώνας. Σας καλώ να ενεργοποιήσετε το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ώστε ο κύριος Φαν να ακούει το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ τόσο πολύ όσο ακούει και το ΕΚΟΦΗΝ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την διακυβέρνηση της Ευρώπης. Δεύτερον, χθες συζητήσαμε για την οδηγία ε, των ε, προσωρινών εποχιακών εργαζομένων με εκπροσώπους της Λιθουανικής ε, Προεδρίας. Ένα μέλος του Συμβουλίου αξιοποίησε την αλλαγή της Προεδρίας για να ξανανοίξει τα θέματα που έχουν να κάνουν με το άρθρο 16 για το οποίο έχουμε εμείς αρμοδιότητα. Θέλουμε να μας βοηθήσετε κυρία Υπουργέ Χθε ήταν πολύ το οικοδομητική η στάση του Συμβουλίου, αλλά ε, πρέπει να το έχετε υπόψη σας γιατί η ίση μεταχείριση είναι κάτι που θα πρέπει να διασφαλιστεί. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ε, κυρία Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Παρακαλώ να είστε ακριβείς. Έξι μέλη της Επιτροπής μας θέλουν να, πάρουν το λόγο. Γι' αυτό καλό είναι να μην καθυστερούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για όλες αυτές τις ερωτήσεις που έθεσαν. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ανρή, Όρη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματά σας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αρρωγής των Περισσότερων Ενδεών. προς την απόσπαση των εργαζομένων είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να προσφέρουμε όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις ε, στους εργαζόμενους όταν έχουν αποσπαστεί και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνέντευξη στο Συμβούλιο και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Είναι λεπτό το ζήτημα, χρειάζεται μεγάλη υπευθυνότητα. Θα κάνουμε το παν για να πετύχουμε συνέντευξη στο Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων βεβαίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προς το Ταμείο Αρρωγής των πιο ενδεών, είναι περίπλοκο το θέμα και αρκετά, με αρκετά προβλήματα. Ε, το ε, επισητιστικό πρόγραμμα στήριξης ε, των πιο φτωχών έχει ολοκληρωθεί, ενώ το Ταμείο θα ενεργοποιηθεί πλήρως του χρόνου. Όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία. Θα κάνουμε το πάντια για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία αυτού του Ταμείου. Ε, ώστε αυτό το ταμείο να λειτουργεί τόσο καλά όσο και το προηγούμενο. Να προσφέρεται συνεχώς βοήθεια, ενίσχυση ε, στους πολίτες που την χρειάζονται περισσότερο. Αναφερθήκατε και στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Είναι μια νέα πρόταση που ε, διαμορφώνουμε αυτή τη στιγμή. Εξ όσο γνωρίζω θα γίνει μία διάσκεψη για το θέμα αυτό τον Οκτώβριο. Η αδήλωτη εργασία είναι ένα φαινόμενο που απαντάται σε όλες τις χώρες. Ε, σε αυτό το πλαίσιο η οικονομικής ανάπτυξης και υψηλών ε, επιπέδων ε, υψηλού επιβιωτικού επίπεδου στα κράτη-μέλη μας ε, προκειμένου να τα διατηρήσουμε αυτά, πρέπει πραγματικά να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία. Ε, στηρίζουμε την πλατφόρμα αυτή και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις. στρέφομαι τώρα προς την κυρία Μπλινκεβίσιωτε. Θέσατε κάποια ερωτήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πρωταρχικά μέτρα αυτό. Επιτρέπει ε, στα κράτη-μέλη να λύσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπινους πόρους. Ε, προβλήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 23,1%. Ενώ ο στόχος είναι το 25% όπως γνωρίζετε. Θέλουμε να πετύχουμε στήριξη και θέλουμε το Ταμείο να καταστεί λειτουργικό από το 2014 και μετά. Όλοι ε, είμαστε υποχρεωμένοι να διαπραγματευτούμε και πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να συνεχίσει να προσφέρει την προστιθέμενη αξία ε, που επιθυμούμε στα κρατη Το δεύτερο σας ερώτημα είχε να κάνει με την ε, προστασία των νέων ε, και με την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδιαφέρονται για την ε, ένταξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων, όλων των κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, αλλά νομίζω ότι ε, υπάρχει παντού. Έχουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Απασχόλησης σε μακροπρόθεσμη βάση, ε, σε βάθος χρόνου. Εκεί μπαίνουν και οι νέοι, αλλά και τα άτομα με αναπηρίες και οι γυναίκες και ο πληθυσμός της υπαίθρου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα ε, εξαιρετικά λεπτό που έχει να κάνει με τις ευαισθησίες πολλών και χρειάζεται απαραίτητη προσοχή. Υπάρχει η αρχή της διαβίου μάθησης. Ε, αυτήν πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε σε σχέση ε, με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι χάνουν τη δουλειά τους. Μιλήσατε άλλωστε για την ποσόστοση υπέρ των γυναικών και για την πρόταση που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα αφορά πολλά κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι η ένταξη των γυναικών σε επιχειρηματικές ομάδες, στον επιχειρηματικό κόσμο, ε, σε πάρα πολλές δουλειές, ε, είναι μια παρουσία αυτή που δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Ε, θέλουμε να πετύχουμε συνένεση. Είπατε ότι επιθυμείτε τη συνένεση και χαίρομαι ιδιαίτερω γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε ε, να βρούμε ευνοϊκές λύσεις στον τομέα αυτό. Κύρια Χόκκινς τώρα, έρχομαι σε εσά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Μας θέσατε ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, για την ανεργία των νέων, για την κοινωνική και εργασιακή διάσταση ε, της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα ξεκινήσω με το Ταμείο ε, Προσαρμογής και Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Όλα τα κράτη-μέλη θέλουν αυτό το Ταμείο να είναι λειτουργικό και να ξεκινήσει ε, τη δραστηριότητά του από το 2014 και μετά. Και πολλές χώρες αξιοποιούν τα κονδύλια του και θα τα αξιοποιήσουν, όπως και η Λιθουανία άλλωστε, η οποία ε, αξιοποίησε τα κονδύλια αυτού του ταμείου πέντε φορές στο παρελθόν. Ε, ξεκινούμε τις τριμερείς διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Όσον αφορά την ενεργεία των νέων, η Ιρλανδία έχει εξασφαλίσει καλά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε τα αποτελέσματα αυτά ικανοποιητικά. για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν πιο σωστή εγγύηση για τους νέους. Τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν χορηγηθεί, αποτελούν ένα καλό αποτέλεσμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν χάρη σε αυτό οι, τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τις συνέπειες της ε, ανεργίας των νέων. Ένα άλλο ζήτημα που είναι η ε, ενσωμάτωση των νέων στην ε, αγορά εργασίας και που χρειάζεται πάλι συνεργασία. Ε, η, αλία, η συνεταιρική αυτή σχέση λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε θα επέτρεπε στους νέους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ε, προσόντα, τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να βρουν μια θέση εργασίας. Θέλω επίση να σημειώσω ότι στην Ευρώπη έχουμε πολλούς νέους που δεν έχουν, ε, δεν είναι εγγεγραμμένοι ούτε σε μαθησιακή διαδικασία, ούτε σε κατάρτιση. Εμείς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Είναι άλλωστε κομμάτι της πολιτικής μας για την νεολαία. Αυτά είχα να πω προς το παρόν και για την κυρία Ζουβέσκα. Θα ήθελα να επανέλθω. Για να πω ότι το θέμα είναι περίπλοκο. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές εμπειρίες και θα πρέπει να επιτύχουμε μια συνένεση ξεκινώντας με τις επιχειρηματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω δε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις στα άρθρα 9 και 10 κυρίως, όπου είναι και τα πιο δύσκολα θέματα για τις κοινωνικές επενδύσεις. Πρόκειται, πιστεύουμε, για ένα στατικό τμήμα της ε, κοινωνικής διάστασης. Και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα συμβούλιο απασχόλησης όπου θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και την επένδυση στην νεολαία. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, πιστεύω, για τα κράτη-μέλη στο σύνολό τους. Πρέπει να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Και πρέπει να επιλύσουμε διάφορα θέματα κοινωνικά, διάφορα προβλήματα. Για τον κύριο Σέρκας, Δεν θα επαναλάβω τίποτα. Από αυτά που έχουν ήδη υποθεί είναι προφανές ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. και να αξιοποιήσουμε το μέσο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Το άλλο ερώτημα. που σχετιζόταν με τους κοινωνικούς εταίρους. Πιστεύουμε Πιστεύουμε ότι κάθε κοινωνική δραστηριότητα η οποία, κάθε επένδυση ε, κοινωνική είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ. Sorry, Ο Στίβεν Hughes και μετά ο Τόμας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα επανέλθω στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και συγγνώμη γι' αυτό, άκουσα τις εξηγήσεις σας. Θέλουμε να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και τρίλογοι μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού εγκρίνεται την κοινή θέση. Απλά Έχετε βάλει μια ημερομηνία για την έγκριση της κοινή θέση ή παρά είναι φιλόδοξο. Δεύτερον, θέσατε, αναφέρετε μεταξύ των προτεραιοτήτων σας την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Δεν αναφερθήκατε ωστόσο, εκτός αν έκανα λάθος, για την νέα στρατηγική, για την υγιεινή και ασφάλεια στην προστασία των εργαζομένων. Μας ε, λυπεί το ότι η Επιτροπή συνεχίζει να καθυστερεί τη δημοσίευση μια νέα στρατηγική υγιεινή και ασφάλεια έχει καθυστερήσει και είναι πολύ σημαντικό να το προχωρήσετε. Επίση, δεν αναφέρεται, το, το ότι δεν το αναφέρετε με ανησυχεί, δεν το αναφέρετε γιατί πιστεύετε ότι θα υπάρξει τίποτα από πλευρά επιτροπή πριν το τέλο τη Προεδρία σα, Αν ναι, θα ελπίζω ότι ω Προεδρία θα ασκήσετε πίεση στην Κομισιό να προωθήσει, να επιταχύνει την δημοσίευση του κειμένου αυτού. Μια τελευταία ερώτηση. Το έθεσε και ο κύριος Σέρκα την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Τονίσετε ότι είναι σημαντική προτεραιότητα για την Προεδρία σας. Εξετάζετε το ενδεχόμενο να κάνετε ένα κοινό συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ΕΠΣΚΟ για να συζητήσετε την, την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η κοινωνική διάσταση θα παραμείνει στο περιθώριο. Τόμασικ και μετά ο Ρίτσαρντ Χάουιτ. Είπατε κύριε Υπουργέ ότι θα καταπολεμήσετε την φαιή οικονομία. Την, όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα με, τη, με την μαύρη οικονομία, με, με την παραοικονομία. Τι θα κάνετε ακριβώς. Ευχαριστώ. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και σύντονη. Ο κύριος Χάουιτ. Και μετά η Ελίζαμπετ Σφέλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και πολύ καλή επιτυχία εύχομαι στην Προεδρεύουσα και εγώ από πλευρά μου. Ένα σχόλιο, μια ερώτηση. Το πρώτο. Εγώ ως Βρετανός μπορώ να σας πω ότι πολλοί συμπατριώτες μου υποστηρίζουν την, ε, τον κανονισμό για την επιστηστική βοήθεια που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και ίσως να μην ε, υποστηρίξουν οι επίσημοι εκπρόσωποι του λαού μας στο Συμβούλιο. Ήθελα να σας το επισημάνω αυτό για να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις που ε, προσπαθούν να δώσουν βοήθεια και ενίσχυση στοχού στην ε, Βρετανία και οι από αυτές ε, υποστηρίζουν ε, τον κανονισμό. Επίσης για την οδηγία για την απόσπαση, εκεί που θα ζητείτε από τις επιχειρήσεις ακροθυγώς μάλλον να καταθέτουν ε, στοιχεία. Αλλά εν περιπτώσει αυτό θεώρησε ο κύριος Μπαρνιέ κατάλληλο. Να καταθέτουν στοιχεία ως προς τις... Ε, την κοινωνική διάσταση της συμπεριφορά των επιχειρησιών τους, ανθρώπινα δικαιώματα, διαφάνεια, διαφθορά και το καθεξής. Είναι κάτι το οποίο έχει μια αλφα ιστορία ως προσπάθεια και εγώ στην Επιτροπή μας αλλά και στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων έχω παρακολουθήσει το θέμα αυτό και οι περισσότεροι συνάδελφοι επίσης. Ε, είχαν υποστηρίξει τον έγινε ψηφοφορία. Περίπου τους 600 βουλευτές είχαν υποστηρίξει το νομοθέτημα αυτό. Ενώ στο Συμβούλιο η Δανία, η Γαλλία, οι κάτω χώρες, η Βρετανία, πατρίδα μου που επέκρινα μόλις τώρα, αλλά από ό,τι ε, μαθαίνω τώρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα προς την πρόταση όπως έχει προχωρήσει. Ε, θα την υποστηρίζαν λοιπόν. Και έτσι όταν μιλούμε για εταιρική ευθύνη και κοινωνική ανάκαμψη ε, και οικονομική ανάκαμψη ε, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό το νομοθέτημα. Άλλωστε και ο Επίτροπος Σάντορ φαίνεται να το προωθεί. Η Προεδρία σας ξέρω ότι δεν ήταν αρκετά ενημερωμένη για το θέμα αυτό και σας είχα επικρίνει στην αρχή. Ίσως χρειαστήκατε περισσότερο χρόνο. Πάντως ε, τώρα φαίνεται να έχετε κάνει κάποιες προκατακτικές συζητήσεις με τα άλλα κράτη-μέλη και ίσως διαπιστώνετε κι εσείς ότι μπορεί να, να ολοκληρωθεί το ζήτημα αυτό, η εξετασία του ζητήματο αυτού και να ληφθούν οι αποφάσει. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία πιο λεπτομερή, για τις προκατακτικές επαφέ. Κυρία Σρότερ, μετά ο κύριος Κρίστινσεν. Ευχαριστώ. Δύο στόμες ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις, κάποια ερωτηματικά που είχα μάλλον έχουν ήδη απαντηθεί, θα τα επαναλάβω. Άλλωστε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και διμερώς για το κοινωνικό πακέτο, για το πακέτο των κοινωνικών επενδύσεων ε, στην απάντηση που είχατε δώσει στις ερωτήσεις μου. Είχατε παραμείνει πολύ γενικόλογοι. Είχατε πει ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε στα παιδιά και ότι ε, μελετάτε κάποια μέτρα κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ γενικόλογα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εάν, πιστεύετε ότι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων είναι προτάσεις που μπορείτε να μεταφέρετε και να υποβάλλετε στο Συμβούλιο. Ε, το δεύτερο θέμα που επίσης δεν αγγίξατε καθόλου αυτή τη φορά, πάλι νομοθετικό ζήτημα για τα διάφορα νομοθετικά ζητήματα που έχουμε να χειριστούμε, ε, η οδηγία για την πολέμηση των διακρίσεων, ένα ζήτημα για το οποίο έχουν αγωνιστεί πολλές προεδρίες, πρέπει να είστε η ένατη ή η δέκατη, ε, που προσπαθεί να βρει μια λύση. Τι μπορείτε λοιπόν να σκεφτείτε εσείς, τι είδους λύσεις μπορείτε να προτείνετε προκειμένου να συμφωνήσει στο Συμβούλιο για την οδηγία αυτή. Όλε Κρίστενσεν. Όλε Κρίστενσεν και μετά η Ευρύν Ρέγνερ. Όλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Υπουργέ για την παρουσίασή σας και ότι και κάθε καλύτερο με τη δουλειά σας. Ξέρετε νομίζω ότι τον, την άνοιση του 2012 οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στον τομέα των κομμωτών συμφώνησαν να προστατεύουν τους κομμωτές από χημικές ουσίες που περιέχονται στις χρωστικές ε, βαφές μαλλιών. Ποια Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό, υπάρχει καμία πιθανότητα αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα και καλή πρόταση να προχωρήσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευλίν Ρέγνερ. Εύλιν Ρέγνερ. Και μετά η κυρία Παπαδοπούλου. Thank you very much. The topic youth unemployment was already mentioned. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκε το θέμα ανεργία νέων. Σήμερα υπερψηφίσαμε ένα σχετικό ψήφισμα και παραπέμπω σε μία παράγραφο που βλέπω στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Πείτε μας λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για την βελτίωση της συνεργασίας των υπηρεσιών δημόσιας αποσχόλησης για να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Τι προγραμματίζετε πιο λεπτομεριακά θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου και μετά θα σου πω και εγώ δύο λόγια. ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στη Λιθουανική Προεδρία κάθε επιτυχία γιατί αναλαμβάνεται σε μια δύσκολη περίοδο. Ήδη και η προηγούμενη Προεδρία, η Ιρλανδική, και πριν η Κυπριακή Προεδρία είχαν θέσει πανομοιότυπους στόχους και δεν βλέπω στις εξαγγελίες τίποτε διαφορετικό. Ο στόχος είναι η πάνταξη της ανεργίας των νέων, δεν ακούω πρακτικά μέτρα, τα 6 δισεκατομμύρια είναι πολύ λίγα που ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό και το ερώτημά μου είναι το εξής πρακτικά μέτρα για την ανεργία των νέων γιατί σήμερα υπάρχει διαρροή εγκεφάλων ε, για τους νέους με πολλά προσόντα από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε άλλες χώρες. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος βιώνουν διαρροή εγκεφάλων ανάμεσα στους νέους. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη. Αναλαμβάνεται λίγους μήνες πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές. Ο ευρωσκεπτικισμός αυξάνεται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι το κοινωνικό κράτος συρρυκνώνεται η ανεργία των νέων καλπάζει και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού νιώθουν έντονα την κοινωνική πίεση από τις αποφάσεις και της τρόικας και τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας. θα ήθελα να δω έμπραχτα τι σκοπεύετε να κάνετε σαν υπουργό ακριβώς λίγους μήνες μετά τις επόμενες ευρωεκλογές για να ξαναχτιστεί εμπιστοσύνη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και των νέων στην ιδέα της ευρωπαϊκής ένωσης σε μια εποχή έντονης κρίσης οικονομικής αλλά κυρίως κρίσης αξιών. Ευχαριστώ. αλλά έχει κλείσει ο κατάλογος των Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομη θα είμαι. Καλώς ήλθατε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ως εισηγήτρια για το Ταμείο Βοήθειας ε, για τους ε, πλέον ενδεείς, θέλω να μου διευκρινίσετε δύο-τρία θέματα. Πρώτον, όπως ξέρετε, και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια Πέρασε ένα ισχυρό μήνυμα ότι πρώτον η χρηματοδότηση για τους φτωχότερους πρέπει να ενισχυθεί και να απευθύνεται στους φτωχότερους και ότι ο προϋπολογισμός των 2,5 δις δεν είναι επαρκής και πρέπει να αυξηθεί στα 3,5 δις. Καταλαβαίνω ότι η απόφαση του Συμβουλίου δέχθηκε τα 2,5 δις για τους φτωχότερους και επιπλέον ένα δις που θα προσθεθεί σε αυτό. Εν ώψη της απόφασης του Συμβουλίου, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει αναστέλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο, πού είναι τα εμπόδια, πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν οι τρεις μερίς διάλογοι για το θέμα αυτό και να συμφωνήσω με τον κύριο Χάουιτ Υπάρχουν χώρες που δεν μετέχουν αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μετάσχουν. Και να τονίσω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Έχουμε μια προεκλογική εκστρατεία το χειμώνα και θα πρέπει να μια περίοδο εν μεσούς, μεσούντος του χειμώνα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πλέον ενδεείς. Υπάρχει επίγον, επίγουσα, ανάγκη επίγουσα αντιμετώπισης του θέματος. Και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα κύριε Υπουργέ για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων μας είπατε ότι ήταν σκληρές οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου τα άρθρα 9 και 12 αυτό συμβεί, σημαίνει ότι για το άρθρο 3 υπάρχει συμφωνία οπότε σε μια τέτοια περίπτωση προς τα πού υπάρχει συμφωνία. Ο Ταβαωρή είπε ότι το κείμενο ήταν ένα κείμενο όπου η απουσία πρόοδου δεν απειλούσε την ασφάλεια δικαίου. Δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι. Για πολλούς λόγους. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου έδειξαν ότι είναι ουσιαστικό, ουσιαστική σημασία να διορθώσουμε τον τρόπο ερμηνείας της υλοποίησης της οδηγίας πέραν της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται, που μετακινούνται, ξέρετε κι εσείς γιατί μετέχετε συζητήσει στο Συμβούλιο, η ευαισθησία για το μέλλον της οδηγίας σε πολλά κράτη-μέλη είναι μεγάλη. Οι συνθήκες υλοποίηση της οδηγίας αυτής θεωρείται ως εμπροσθοφυλακή της δημιουργίας ενός κοινωνικού dumping και της αποσύνθεσης του εργατικού δικαίου στις περισσότερες χώρες μέλη. Άρα υπάρχει ανάγκη επίγουσας λύσης για την εγγύηση νέων. Το αναφέρατε. Σας εφιστώ την προσοχή στη θέση του Κοινοβουλίου, θέση που θεωρούμε πολύ σημαντική. Το Συμβούλιο το Φεβρουάριο στο ΕΠΣΚΟ, κάτι που επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο στο Συμβούλιο Γεωργίας, την σημασία αυτής της εγγύησης για τους νέους. Και το ίδιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο. Έχω ωστόσο την εντύπωση ότι στο Συμβούλιο δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα του θέματος. Διότι αν πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντική η εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να καταγραφεί σαφώς ότι ο προπολογισμό του, του Κοινωνικού Ταμείου επιτρέπει τη χρηματοδότηση την διαδικασία αυτή. Αυτή τη στιγμή ωστόσο η οδηγία, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περιέχει αβεβαιότητες. Ο κανονισμός εν γέννη μπορεί να βοηθήσει το μηχανισμό εγγύησης νέων αφενός, από την άλλη ωστόσο η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, τα 6 συν 2 δις, πρέπει να μπορέσει να υποστηρίξει την εγγύηση νέων. Τρίτο σημείο αναφέρατε το έγγραφο που υπεγράφει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Επιτροπής και του Συμβουλίου στις 2 Ιουλίου. Θα το συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους στο τέλος της συνάντησής μας σήμερα. Τελευταίο θέμα για το Ταμείο για τη Φτώχεια. Είπατε ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν το είπε και ένα συνάδελφο. Από πλευρά Κοινοβουλίου, ειλικρινά σα το λέω, ελπίζουμε ότι μετά από δύο συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με συμπεράσματα που επαναλήφθηκαν στο Συμβούλιο 27-28 Ιουνίου που είπαν πέντε δις εκ των οποίων 2,5 υποχρεωτικά θα υπάρξει η υλοποίηση προσανατολισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις επί της ουσίας του θέματος, γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε διέξοδο. Πάντως ευχαριστούμε που μας ανησυχήσατε, που μας προειδοποιήσατε. Έχουμε και εδώ λόγους να ανησυχούμε. Πάντως οι πρακτικές εργασίες του Συμβούλιο θα πρέπει να παρακολουθούν, νομίζω το ξέρετε αυτό, αρμονικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε στις τελευταίες ε, παρατηρήσεις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών. Ευχαριστώ. Για τις ερωτήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικές και για σας και για μας. Και ξεκινώ με την ερώτηση του Στίβεν Χιούς για την υγεία και ασφάλεια καταρχάς. Δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί πρώτα στην Επιτροπή. Όταν έρθει η ώρα θα το υποβάλουμε στο Συμβούλιο και αν χρειαστεί θα ξεκινήσει η συζήτηση για το σημαντικό σου και ευαίσθητο αυτό θέμα. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε για τον Νοέμβριο. Δεύτερο θέμα. Κοινωνική διάσταση. Όπως είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι πολύ σημαντική η κοινωνική διάσταση. Οι μελέτες δείχνουν ότι η οικονομική και κοινωνική τομείς ε, είναι σχετική και μπορεί να διαταραχθεί η κοινωνική σταθερότητα. Άρα λοιπόν, ε, ναι μεν είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας, αλλά χρειάζεται κάποια στιγμή να δούμε ότι με, μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτών θα φέρουν αρκετά πλονεκτήματα και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και τη δυνατότητα να ε, προβλέψουμε ενδεχομένες ε, ανισορροπίες για να λάβουμε μέτρα εγκαίρως. Δύο επιτροπές ασχολήθηκαν με την ε, κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση έχουν δύο ε, συστήματα παρακολούθησης, επιτήρησης. Για να επιτευχθεί πρόοδο στον τομέα αυτόν, θα πρέπει να Έχουμε κοινωνικού δείκτες, Πίνακε αποτελεσμάτων, scoreboard του ονομάζουμε, για την κοινωνική κατάσταση και την απασχόληση. Και έχουμε στοιχεία. Έχουμε επισημάνει τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να είναι ένα επιπλέον βάρος, αλλά θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, παραδείγματι, για να τα συλλέξουμε. στην επιτήρηση και το συντονισμό, ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά ως προς την, κοινωνική, ως προς την κοινωνική πτυχή για τους αποσπασμένους. Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ τον Οκτώβριο θα επιδιώξει να προχωρήσει στη λήψη μιας απόφασης. Και αυτή είναι η τελευταία πάτηση που σας δώσω. Και θα είχα και μια πολύ άμεση απάντηση για το πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις στην απασχόληση. Ανεργία λοιπόν υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος. Και μεμονωμένα το κάθε κράτος ή υπηρεσία δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ενέργεια. Έτσι λοιπόν χρειάζεται συμμετοχή και κοινωνικών εταίρων και άλλων θεσμών που θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί ο τομέας και η πρόταση αυτή μπορεί να επιτρέψει να αναγίνει μια ανάλυση κατάσταση στα κράτη-μέλη και να ρυφθούν αποφάσεις E, e, και επίση, τον Οκτώβριο πιστεύω θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων στη διάσκεψη που οργανώνουμε. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Αυτά για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση. Για τον κύριο Χάουιτ έχω να πω τα Μιλήσατε για το Ταμείο και τους πιο δύναμους οικονομικά. Όπως ε, προνέφερε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το Ταμείο είναι, πιστεύω, μία από τις δυνατότητες να καταπολεμήσουμε τις συνέπειες της ε, φτώχειας. 2,5 δισεκατομμύρια αντί για 3,5 που είχε στο Κοινοβούλιο έχουν προβλεφθεί για το Ταμείο. Και το 1 εκατομμύριο που λείπει θα πρέπει να συζητηθεί από πού μπορούμε να το βρούμε. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ζητήσουν και από το εθνικό επίπεδο λύσει στα προβλήματα τη φτώχεια. Ο κύριος Χάουτ μίλησε και για κοινωνική ευθύνη επίση. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητο σε όλους τους τομείς. Και καθώς το θέμα αυτό είναι εγγράφητο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των αρμοδίων για τα οικονομικά, αν εμείς ασχολούμαστε με την απασχόληση περισσότερο, την ερώτηση σας θα την, την παρατήρησή σας για τη σημασία των κοινωνικών ατέρων θα την παραπέμψω στον άλλο συνάδελφο Υπουργό των Οικονομικών. atsakyti dėl socialinių investicijų paketo, kad... Για να απαντήσω τώρα στην κυρία Σρέντερ για το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Όπως είπα προηγουμένω. είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα η επένδυση στα παιδιά που αναφέρατε. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Οι δυνατότητε να πάνε στο σχολείο, να σπουδάσουν, να ενσωματωθούν σε κοινωνικές δραστηριότητες, μπορεί να τους βοηθήσουν, να βοηθήσουν να έχουν μια σαφή εικόνα μέσα στην κοινωνία, ε, παρουσίαση μέσα στην κοινωνία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσει να εκπαιδευτεί η νέα γενιά και να έχουμε μέσα και εργαλεία για να βοηθήσουμε τους νέους να φτάσουν, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην, στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, να έχουν ευκαιρίες εν για να ενταχθούν στην κοινωνία. για τη δεύτερη ερώτησή σας. Η οδηγία κατά των διακρίσεων. Είμαι σίγουρη ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, ευχαριστούμε την Ιρλανδική Προεδρία που έκανε τεράστια πρόοδο στον τομέα. Το πρόβλημα είναι ότι στο άρθρο 19 χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη και περιμένουμε να υπάρξει συνένεση. Στην κυρία Κρίστενσεν. Στον κύριο Κρίστενσεν. Συγγνώμη που έφερε την ερώτηση για τους κομοτές και τις κομμότριες. Και το ότι έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες από τις βαφές μαλλιών. Η Επιτροπή κάνει μια μελέτη αντικτύπου και φαντάζομαι ότι θα υποβάλω μια σχετική πρόταση το στομό το δυνατό. Οπότε θα εξετάσουμε το θέμα μεταγενέστερα. Ίσως να υπάρξει και κάποια σχετική απόφαση. Για την κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για τις υπηρεσίες απασχόλησης. Πιστεύω ότι όσο ισχυρότερες είναι οι υπηρεσίες απασχόλησης σε κάθε κράτος μέλος, τόσο ευκολότερα θα ενταχθεί ο νέος στην αγορά εργασία. Είναι σημαντικό λοιπόν οι υπηρεσίε απασχόλησης να συνεργάζονται μεταξύ, οι υπηρεσίε απασχόλησης κάθε κράτους μέσα να συνεργάζονται μεταξύ τους δηλαδή. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και να αποκτούν διάφορες και διαφορετικές εμπειρίες. Το EURES το δίκτυο γιούδες και το δίκτυο των υπηρεσιών έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν. Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για την βελτίωση της δομής λειτουργίας των οργανισμών απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Πιστεύουμε ότι θα δουλέψουμε πάνω στο κείμενο αυτό και θα συνεχίσουμε τη δουλειά. για την ερώτηση της κυρίας Παπαδοπούλου και της Προέδρου. για την απασχόληση των νέων και το πρόγραμμα εγγύησης ε, για τους νέους. Σε ό,τι αφορά την εγγύηση νέων, με χαρά διαπιστώσαμε την πρόοδο που επιτέχθηκε επί Ιρλανδικής Προεδρίας. Αυτό ωστόσο είναι μία μόνο από τις ευκαιρίες να βελτιώσουμε την αποσχόληση μεταξύ των νέων. Πιστεύουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να προβάλλει πόρους ίσως και του κοινωνικού ταμείου για να επιταχύνει την απασχόληση μεταξύ των νέων. Όπως είπα, υπογράψαμε την, το επίδομα μαθητείας φέτος τον Ιούλιο, που θα πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα που θα βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν τα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν περισσότερο στην αγορά εργασία. Και πάλι ανέφερα το πρόβλημα των αναγκών είναι σημαντικό να κάνουμε τους νέους πιο δραστήριους και τα τρία αυτά ντοσιέ είναι μεταξύ των βασικών μας προτεραιοτήτων. Η εγγύηση νέων θα συζητηθεί στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ τον Οκτώβριο και θα καλέσουμε τους υπουργούς να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για να διευκολύνουν την υλοποίηση της εγγύησης νέων. Θα διασφαλίσουμε ότι τα ταμεία, οι πόροι για την εγγύηση νέων θα χρησιμοποιούνται ιδίω στην αρχική περίοδο, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό. Τελευταίο για την κυρία Κοστέλο για τη μείωση της φτώχειας. Προφανώς μας ικανοποιεί η ύπαρξη του Ταμείου. Klausite konkrečiai, tai e, Liepos 17 dieną bus pradėtos dėrybos koreperų lygmenį. Τώρα, για την ερώτησή σας. Οι διαπραγματεύσει στην Κορεπέρ θα ξεκινήσουν 17 Ιουλίου. Θα είναι ένα από τα βήματα, ένα από τα αρχικά βήματα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε Ελπίζουμε κυρία Υπουργέ ότι από αυτή την ανταλλαγή απόψεων αποκομίσατε κάποιες βασικές εντυπώσεις για τις προτεραιότητες των μελών της Επιτροπής μας. Πολλά από αυτά που μας είπατε δείχνουν ότι είναι και προτεραιότητες του Συμβουλίου, ωστόσο κάθε θεσμικό όργανο έχει τη δική του οπτική γωνία. Ως προς το θέμα των κομωτών, θα πρέπει να το προσέξει η Λιθουανική Προεδρία, πιστεύω. Δεν έχει τεθεί επιτάπητος επισήμως, διότι ε, δεν έχει ε, συσταθεί Επιτροπή. Ωστόσο, είναι μια παλαιά συμφωνία αυτή μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και συνεχώς όλοι ε, τίθενται υπέρ ε, του κοινωνικού διαλόγου. Είναι μια συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Εμείς το είχαμε θέσει το θέμα στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τον περασμένο Οκτώβριο και από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει το θέμα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να επιταχυθεί κάπως η διαδικασία, να φανεί ότι τα λαμβάνει θετικά υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά θετικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ε, εκεί χωλαίνει κάπως το πράγμα και είναι κρίμα. Και είναι σημαντικό από τη στιγμή που ξεκινάτε τώρα την ε, Προεδρία σας να σας το επισημάνουμε. Ε, σας ευχαριστώ θερμά εξ ονόματος όλων των μέλων της Επιτροπής μας. Θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη όταν θα έχετε την τιμή να μας υποδεχθείτε στους στο πλαίσιο της ε, συνεδρίασης ΕΠΣΚΟ. Εν τω μεταξύ σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, Προεδρία σας. Bien. Euh... Sans plus attendre, je vous propose euh, de revenir à notre ordre du jour. Λοιπόν, σας προτείνω να επανέλθουμε στην ημερήσια διάταξη και να πάμε στο σημείο 16, ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά Απόβλητα στο Περιβάλλον. Είχαμε εξετάσει τη γνωμοδότηση της Τζιν Λάμπερτ. Είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή, ε, την αρμόδια την Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία ο αρμόδιος εισηγητής είναι ο κύριος Πρόντι. Ε, δίνω το λόγο στην κυρία Λάμπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε κι εσείς, είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, διότι θελήσαμε να ανταποκριθούμε, να αντιδράσουμε στην πράσινη βίβλο που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα για τη στρατηγική διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Βεβαίω η περιβαλλοντική διάσταση είναι εξαιρετικά παρούσα, αλλά αξίζει το θέμα να το δούμε και ε, στο πλαίσιο της πολιτικής ε, αποδοτικότητας των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 60 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων παράγουμε βάσει των εκτιμήσεων που επικρατούν στην Ευρώπη κάθε χρόνο και 15% του πλαστικού μας καταλήγει σε χωματαερές, κυρίως υλικό συσκευασίες, 12 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου δηλαδή. Είναι περιβαλλοντικό το πρόβλημα. Πολύ, πολλά από αυτά τα πλαστικά απόβλητα δεν αποσυντήθεται. Πολλοί πιστεύουν ότι αποσυντήθεται, αλλά δεν ισχύει. Και ένα τελικό 15 ε, ε, καταλήγει στην ενεργειακή ανα, ε, ανάκτηση, ε, καύση και στην ανακύκλωση βέβαια. Ανακυκλώνουμε λίγο πάνω από το 25% ε, των πλαστικών αποβλήτων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαφορές είναι τεράστιες βέβαια μεταξύ των κρατών μελών. Κάποιοι ανακτούν σχεδόν το 90% των πλαστικών αποβλήτων, ενώ άλλοι ε, θάβουν ε, σχεδόν το 90% των πλαστικών τους αποβλήτων. Και μάλιστα πολύ συχνά η συλλογή των πλαστικών αποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο είναι πολύ πιο αποτελεσματική σε κάποια κρατημέλη από ό,τι σε άλλα. 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο της ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξάγουμε αυτή τη στιγμή και πολλά ε, πλαστικά απόβλητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, εξάγει τα πολλά πλαστικά απόβλητα του στην Κίνα και στην Άπο Ανατολή και έχουμε δει και αλλαγές στην νομοθεσία της Κίνας αυτή τη στιγμή. Ε, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προκλήσεις στην Ευρώπη για εμάς και πολλοί από εμά ε, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την άρνηση που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δεν θα θέλουν να υποδεχθούν τα μη ε, ε απόβλητα στα οποία δεν έχει γίνει διαλογή, ανακύκλωση και το καθεξής. Τώρα, με την ανακύκλωση έχουμε ένα μείγμα ε, δουλειάς υψηλής τεχνολογίας, αν επισκεφτείτε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης ε, γυάλινων φιαλών για παράδειγμα, θα δείτε αμέσως, θα διαπιστώσετε αμέσως ότι ορισμένοι εργάτες είναι ανειδίκευτοι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ε, εργαζόνται εκεί ε, άνθρωποι με υψηλά προσόντα και ε, οι απαιτήσει από πλευράς τεχνολογίας είναι εξαιρετικά υψηλές. Απαιτείται προηγμένη τεχνολογία για όλα αυτά. Όλα αυτές είναι κάποιες βασικές παρατηρήσεις που θέλω να κάνω για τη συζήτηση. Προφανώς ένα από τα βασικά ζητήματα έχει να κάνει με την αξιολόγηση αντικτύπου των πρωτοβουλειών για την πολιτική για το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ποιες ευκαιρίες έχουμε στην πολιτική για το περιβάλλον να ενισχύσουμε την πολιτική της απασχόλησης ε, και της αγοράς εργασίας. Θέλουμε μια ανάκαμψη οικονομική, η οποία να είναι πλούσια σε δουλειές και πλούσια σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά συντεριάζουν με τη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και για μια βιώσιμη, αηφόρο οικονομία έχουμε και τους στόχους στην οδηγία πλαίσιο και την οδηγία για τη συσκευασία ε, αποβλήτων ε, και εκεί δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται το δυναμικό αυτό των οδηγιών. Η ανακύκλωση είναι ένας κλάδος υψηλής εντάσεως εργασίας ούτως ή άλλως και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πολλές από τις καινοτομίες που έχουν υπάρξει στον τομέα των πλαστικών ε, έχουν επηρεάσει άμεσα και την ε, ε, επαναχρήση, την εκ νέου χρήση και θα πρέπει να ε, δούμε προσεκτικά και το, τη διάσταση της ασφάλειας. Δημιουργούνται νέα προϊόντα γεμάτα νανοτεχνολογία. Έχουμε όλο και περισσότερο καλλιντικά που έχουν μικρά σωματίδια από πλαστικό, στις μάσκες για παράδειγμα ε, προσώπου, ε, οι οποίες καθαρίζουν τους σπόρους ή ε, κρέμες ε, για να φαίνεται λαμπερή επιδερμίδα έχουν και ε, σωματίδια πλαστικού μέσα. Υπάρχει δηλαδή και μια διάσταση της υγείας σε όλα αυτά και που θα πρέπει να δούμε και τέλος θέλω να αναφερθώ στην κατάρτιση και στα προσόντα, στις δεξιότητες στον τομέα αυτό. Να ε, διασφαλίσουμε ότι και αυτά τα θέματα τα προχωρούμε. Δηλαδή δεξιότητες, κατάρτιση, εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη νέα νομοθεσία. Ε, σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας χρειάζεται και ε, το κενό παραμένει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και μεγάλο. Δηλαδή υστερούμε σε προσόντα και δεξιοτεχνίες. Η απαραίτητη και η κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση είναι αυτό που κάνει όλους να καταλάβουν τελικά γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η δουλειά. Και πρέπει να αλλάξει και η αντίληψη που έχουμε για το κοινωνικό καθεστώς ε, όλων αυτών που εργάζονται στην ανακύκλωση ε, και σε αυτούς τους τομείς. Θεωρείται ότι είναι μια δουλειά που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε, των αντίον. Ε, και μάλιστα είναι μια πολύ σημαντική δουλειά Ειδικά αν σκεφτεί κανεί τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ανακύκλωση και όλα αυτά ε, τα πετάγαμε έτσι ελεύθερα στην ατμόσφαιρα ή στη φύση. Εν πάση περιπτώσει, η ε, τροπολογία. Ε, ε, και το κείμενο περιλαμβάνουν όλες αυτές ε, τις παρατηρήσεις που δεν ε, μπόρεσα να περιλάβω στους αρχικούς 1500 χαρακτήρες. Περιμένουμε και το επόμενο στάδιο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου παρακαλώ. Thank you, Chair. I am the Ευχαριστώ. Είμαι η συγγήτρια Σκιώδης από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε νομοδότηση αυτή. Είναι ευπρόσδεκτη φυσικά η οδηγία για, ε, για τα απόβλητα. Έχει κάνει μια καλή γνωμοδότηση κυρία Λάμπερτ. Διατυπωμένη σωστά, καλυπτεί τα περισσότερα θέματα που μας απασχολούν. Θα θέλαμε απλώ να ενισχύσουμε το κείμενο με την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις κοινωνικές, ε, τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας της στρατηγικής γιατί για να επιτύχουμε μια τέτοια στρατηγική και τη σχετική ανάπτυξη πρέπει να μιλήσουμε για μια βιώσιμη ποιότητα στις θέσεις εργασίας, στην διαχείριση των αποβλήτων και βέβαια δεν πρέπει να υποτιμούμε και την ε, ιδέα ότι υπάρχει περιθώριο όχι μόνο απασχόλησης, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση που θα μειώσουν την ένταση πόρων σε πρώτη φάση. Στο πρώτο στάδιο προκαταβολικά δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρερ από την ε, Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον είχε έρθει και νωρίτερα, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει τόσο αργά. Μου ζήτησε να σα επιβεβαιώσω ότι το σχέδιο γνωμοδότηση είναι πολύ ε, συμβατό με την ε, πράσινη βίβλο. Μου ζήτησε να σας επιβεβαιώσω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα αυτό. Κύριε Λάμπερτς, ευχαριστώ για τα σχόλια. Περιμένουμε να δούμε και τις τροπολογίες που είμαι σίγουρη ότι θα προσφέρουν κάτι, θα συμπληρώσουν το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Κατάθεση τροπολογιών στις 17 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Με ηλεκτρονική υπογραφή σας υπενθυμίζω, με γιατί έγινε αυτό, αλλά έτσι είναι. 25-26 για να εξετάσουμε τις Σεπτεμβρίου για να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ψηφιακή η υπόγραφη λοιπόν για να κατευθούν οι τροπολογίες 17 Ιουλίου. Εξέταση τροπολογιών 25-26 Σεπτεμβρίου. Και αν το επιτρέπει το χρονικό μας περιθώριο, εξέταση και ψηφοφορία τον Οκτώβριο στη συνεδρίαση την ίδια μέρα για να το αρμόδια καθήλυν. Επιτροπή τον Νοέμβριο και τώρα τελειώνουμε το θέμα αυτό και στο 25 παρακαλώ την ε, κυρία Ζδάνοβα να λάβει το λόγο για να μας μιλήσει για την οργάνωση μιας δημοσκόπησης σχετικής με το εργατικό δυναμικό μέσα στην κοινότητα. Πρόκειται για έκθεση στην οποία η Επιτροπή Προπολογισμών θα γνωμοδοτήσει και η συγκέντρια έχει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση της Επιτροπής είναι τεχνικού χαρακτήρα Οι τροπολογίες μας ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικές αλλά και πολιτικές. Αφορούν πρώτα-πρώτα την αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασία. Το θέσαμε το θέμα αυτό σήμερα στην ερώτηση προς την Λιθουανή Υπουργό Ξέρει ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και εγώ ήμουν υπεύθυνο της στρατηγικής της Ένωσης ε, για την μη διάκριση και διαπίστωσα την έλλειψη πληροφοριών ενημέρωσης. Η πρότασή μας διευρύνει την προαιρετική υποβολή απαντήσεων σε ερωτήσεις προτείνουμε να υπάρξουν προεκτικές ερωτήσει για την εθνοτική ή φυσική ε, η εθνική προέλευση, σεξουαλική ε, γενετήσια, γενετήσιο προσανατολισμό κτλ. Όλα αυτά καλύπτονται και στο άρθρο 4, 1, 2. Προφανώς αναφέρεται ότι ο, ε, ο σεβασμός των στατιστικής εμπιστευτικότητας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων λοιπά. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει την τροπολογία αυτή. Δεύτερον, για διαδικαστικά θέματα που πρέπει να οδηγήσουν στην αντικατάσταση της κανονικής διαδικασίας με εξέταση. Η Επιτροπή προτείνει προτείνει εκτελεστικές πράξεις, εμείς προτείνουμε κατεξουδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 5 και στο τμήμα 2 του άρθρου 4. Η τρίτη πρόταση αφορά τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Έχει και γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και περιλαμβάνουμε μία επιφύλαξη για πραγματική υλοποίηση. Τέλος, η τελευταία μεγάλη τροπολογία αφορά την περίοδο εξουσιοδότησης. Σα είπα ότι προτείνουμε κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Προτείνουμε όχι απεριόριστη διάρκεια, αλλά πενταετούς διάρκεια Περιλαμβάνεται στο άρθρο 7.3 γάμα. Αυτές είναι οι προτάσεις μου, ελπίζω να τις επιταχύνετε και να τις υποστηρίξετε. Η κυρία Ισαΐα και μετά η κυρία Άρκιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις τροπολογίες της. Να ξεκινήσω με τις τροπολογίες ένα και τέσσερα. Καταλαβαίνω ότι η συγκήτρια έχει στόχο να καταπολεμήσει την διάκριση. Δεν συμφωνώ ωστόσο τούτο να γίνει μέσω της ε, έρευνας εργατικού δυναμικού, διότι εκεί περιλαμβάνονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Είναι σημαντικό να απαντούνται. Εάν σε μια τέτοια έρευνα περιλαμβάνουμε ερωτήσεις ευαίσθητου χαρακτήρα όπως εθνοτική προέλευση, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, ε, αναπηρία, κάποιοι μπορεί να πούν ή να σκεφτούν ότι καλό είναι να μην απαντήσουμε καθόλου. Δεν πρέπει λοιπόν να θέσουμε σε κίνδυνο κάτι τέτοιο. Παρότι τα θέματα αυτά είναι σημαντικά, και πρέπει να τα ξέρουμε, δεν πρέπει να γίνεται αυτό στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό συμφωνώ, διαφωνώ, συγγνώμη. Για το πού πρέπει να γίνονται οι ερωτήσεις αυτές, όχι αν πρέπει να γίνονται ή όχι. Το άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω Κάποιες από τις προτάσεις Επιτροπής για τους κανόνες πρέπει να γίνονται με μια σειρά τυπικών διαδικασιών, φερρυπίν, τεχνικού χαρακτήρα. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ε, χρειάζεται κατεξοδότηση πράξης. Τρίτο θέμα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια να υπάρξει πενταετής περίοδο εκχώρησης εξουσιών, ε, κατεξοδότηση πράξεων. Εμείς επιπλέον θέλουμε τρίμηνο για να ελέγξουμε τη χρήση κατεξοδότηση πράξεων και θα υποβάλω μια σχετική τροπολογία. βλέπω στη συνέχιση των εργασιών με τους υπόλοιπους ε, Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την συγκίτρια για την παρουσίασή της. Τεχνικό είναι το θέμα όντως. Και εγώ είχα μια ερώτηση για την τροπολογία 1 και 4. Παρόμοια με αυτή της κυρίας Εσάια Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε αντικειμενικές συγκρίσιμες πληροφορίες επί των οποίων να βασίζουμε τις δράσεις μας. Το ερώτημα είναι, είναι αυτός ο καταλληλότερος τρόπος συλλογής των πληροφοριών αυτών. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαιη. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, δεν έχω πρόβλημα και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Επιτροπής. Φοβάμαι μήπως αυτές οι ευαίσθητες πληροφορίες θέσουν ε, σε κίνδυνο την ακρίβεια των στοιχείων του, της έρευνας εργατικού δυναμικού. Και η ερώτηση προς την Επιτροπή είναι με βάση ποιο στοιχείο εκρίνεται, ε, οι επιλογές ε, των ερωτήσεων. Είπατε επίσης στην Επιτροπή ότι τρεις στόχοι καλύπτονται Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις στόχοι. Υποστηρίζω την εισηγήτρια για την περίοδο εξουσιοδότησης και στο άρθρο 4.2 υπάρχει πρόταση να προχωρήσουμε από εκτελεστικές σε κατεξιοδότηση πράξης. Θα έλεγα οι κανόνες διαμόρφωσης των μεταβλητών είναι τεχνικοί, άρα δεν χρειάζεται κατεξουσιοδότηση, αλλά ο κατάλογος των αρχών που θα διέπουν αυτές τις μεταβλητές μπορεί να περιλαμβάνει και πολιτικά στοιχεία, οπότε ίσως εκεί να πρέπει να εξετάσουμε την εξουσιοδότηση. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η κυρία Κοστέλα όμως εν μεταξύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό, ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό. Υπόθηκε ήδη ότι τα στοιχεία της έρευνας ε, ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη. Αλλά τα top modules ενδιαφέρουν κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώ στην κυρία Χάρκιν και εκφράζω την ανησυχία μου. Οι δείκτες λένε ότι τα modules της στρατηγικής του 2020 είναι ένα στόχος απασχόλησης 75%. Όσοι εγκαταλείπουν το σχολείο να μην ξεπερνούν το 10% και όσοι φτάνουν τα ένα 30% τουλάχιστον να ολοκληρώνει τριτοβάθμια εκπαίδευση. 30 με 35%. Αυτός ο φάκελος ουσιαστικά θα αποτελέσει τη νομική βάση ώστε η Επιτροπή να δώσει επιδοτήσεις σε χωρίς διαγωνισμό. Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές τα στοιχεία μας υστερούν, μερικές φορές δυσκολευόμαστε να έχουμε στοιχεία για την ηλική στέρηση. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ως προς την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση Ένα από τα top modules μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση που θα δώσουμε στους νέους ε, για αυτό το σύστημα. Κάποιες ερωτήσεις τεχνικής φύσης έχω να υποβάλω και όποιες τροπολογίες υποβάλλω θα έχω να κάνουν με τις λεπτομέρειες και όχι με την ουσία. Ε, κάποιος ομιλητής σε σχέση με την τροπολογία υπαρθμών 1 είπε κάτι. Να ρωτήσω λοιπόν την εισηγήτρια. Έχετε τάση αναφορά το ευρύτερο άρθρο 21 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει να κάνει ε, με τις διακρίσεις που θα πρέπει να καταπολεμηθούν βάσει των γενικών χαρακτηριστικών. Είναι ένας τρόπος καταπολέμησης των διακρίσεων. Είναι ένα παράθυρο που αντίγεται δηλαδή. Και, τους, και ως προς την προαιρετική φύση, το optional, ε, στην ε, τροπολογία 4. Μήπως θα πρέπει να το εξετάσει το Συμβούλιο αυτό. Και από εκεί και πέρα, η πρόταση για πλήρη συμμετοχή θα μπορούσε να υπονομεύσει ε, τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να διευκολύνονται τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στα top modules σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε σχέση με το DAC και την τροπολογία 10 και τις κατεξουσιοδότηση πράξης, τι εννοούμε με το tacitly extended, σιωπηλά επεκτείνεται αυτή η περίοδος εξέτασης. Ίσως σχετίζεται με μια περίοδο από 2-5 χρόνια. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με τους κυρώδες εισηγητές ε, και θα υποβάλουμε τις αντίστοιχες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, να σας πω ότι διαβάζατε εξαιρετικά γρήγορο, γρήγορα και αυτό δεν είναι καλό για τη δερμηνία. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν το αντιλήφθηκα προ... νωρίτερα. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να μας πει και για τη Eurostat και όλα αυτά. Όμως εγώ ε, δεν βλέπω ο τίτλος να έχει προσαρμοστεί. Είναι απαξιωμένος, είναι απερχιωμένος. Μιλάει για την κοινότητα δεν θα χρησιμοποιούμε πια τον όρο κοινότητα στα νομοθετικά μας κείμενα, έτσι δεν είναι. Μήπως πρέπει να, διατηρήσουμε το χαρακτηρισμό κοινότητα σε αυτό το νομοθέτημα και αν ναι τότε θα μου εξηγήσετε το γιατί. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι υπεύθυνη για το φάκελο αυτό. Αντικαθεστώ τη συνάδελφο στη γύρω. εξετάζουμε τον κανονισμό αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 1998. Και σκοπός είναι να, προσαρμόσετε, να προσαρμόσουμε αυτό το κανονισμό στο νέο θεσμικό πλαίσιο και να μπορέσει η Επιτροπή ε, ε, να έχει οικονομική ε, συνδρομή. Κάθε χρόνο τα modules τα προσδένουμε στο survey, στην έρευνα και θέλουμε ε, να δίνουμε κάποιες ενισχύσεις στις χώρες. Τρία θέματα έχουν τεθεί στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Πρώτον, το, τα optional valuables. Προτείνουμε δηλαδή να προσθεθούν κάποιες πληροφορίες προαιρετικές για την αναπηρία, για την εθνοτική προέλευση και ούτω καθεξής πολύτιμα στοιχεία. Η έρευνα για το εργασιακό δυναμικό δεν είναι το εργαλείο ε, με το οποίο θα συλλέξουμε τέτοια στοιχεία και τέτοιες πληροφορίες. Σίγουρα θα συμφωνείτε με αυτή την ε, παρατήρηση. Θέλουμε πληροφορίες για την αγορά εργασίας και δεν θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες που να θέτουν ένα αμφιβόλο τις απαντήσεις των ατόμων. Έχουμε άλλη έρευνα για τις αναπηρίες. Εάν σας ενδιαφέρει να έχετε στοιχεία για τις αναπηρίες, έχουμε άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Αλλά για την ηλική στέρηση επίσης ε, έχουμε άλλο εργαλείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Από την άλλη πλευρά, σε μια έρευνα όπου ε, υπάρχουν ερωτώμενοι, αποκρινόμενοι, είναι δύσκολο να συλλέξουμε ε, ε, πληροφορίες για τα πιστεύω, για την εθνοτική προσέλευση. Είναι πολύ λεπτές πληροφορίες και δύσκολα τις συλλέγουμε άμεσα από τους ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, διότι στην τελική ε, μπορεί να μην, πάρουμε και να μην πετύχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Και ως προς την αναπηρία έχουμε ειδικό εργαλείο. Ε, ως προς τις κατεξουσιοδότηση πράξης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέμε εμείς ότι για τον ορισμό των valuables που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο module ή των διαρθρωμένων τέλος πάντων valuables, προτείνουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξη λόγω της ε, τεχνικής φύσης, ε, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά τεχνικά τα ζητήματα αυτά. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε αυτά να τα ρυθμίσουμε με ε, τα εφαρμοστικά μέτρα. Τώρα, ως προς τα θέματα χρηματοδότησης, η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει σαφέστατα ότι δεν είναι αποδεκτό για εμάς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις αυτές, οι, ε, υποτροφίες αν θέλετε, να δίδονται εφάπαξ θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στον κανονισμό. Δηλαδή να δίδονται αυτά τα ποσά με τον πιο κατάλληλο τρόπο κάθε φορά. Ε, και τέθηκε και ένα ερώτημα για το RVT, για τα modules που επιλέγουμε. Τα θέματα συνδέονται πάντοτε με την αγορά εργασίας, ξέρετε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αποφασίζουμε αυτά. Είναι μια μεταβατική περίοδος ε, για την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, για την είσοδό τους. Κάποιες λοιπόν θεματικές ενότητες θα έχουν σίγουρα να κάνουν με θέματα της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Συγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις προς τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή. Έχουμε συναντηθεί βέβαια ήδη με εκπροσώπους και της Eurostat. Έχουμε θέσει τις ερωτήσεις μας, έχουμε λάβει τις απαντήσεις μας, έχουμε συζητήσει τις διάφορες προτάσεις. και για... τις απαντήσεις. Πρώτη αντίδραση, όχι εδώ, αλλά πού. Δεν έχουμε να κάνουμε μια ad hoc. ελέτη. επομένως, ε, το να θέσουμε τα ερωτηματικά σαν να παρουσιάζεται κατά τρόπο ε, εκούσιο ο χάρτης. Δεν ξέρω για διακρίσεις, αλλά έχουμε εξετάσει πολλές δυνατότητες. Δεν αντιτίθεμε, τα, τα σημεία αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα Η έκθεση έφτασε το 2007. Αρχικά είχαμε αντιδράσεις από ορισμένε πολιτικές ομάδες. Ταυτόχρονα όμως τα επεισόδια στις, στα προάστια του Παρισιού αλλά και άλλων πρωτεύουσων. Και η λεγόμενη κρυφή, η συγκεκαλυμμένη διάκριση που προβλήθη εξαιτία αυτών, μας υποχρέωσε να συζητήσουμε θετικά μέτρα για την αποφυγή και την καταπολέμηση των διακρίσεων, Όλοι μιλάμε για εγκάρσια οδηγία. Δεν την έχουμε ακόμα εξασφαλίσει. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενες οι προτάσεις. Θα ήθελα να τις συζητήσουμε. Ως πολιτικοί πρέπει να επιδείξουμε θάρρος για να προχωρήσουμε με τέτοιου είδους προτάσεις. Ιδάλλως δεν έχει νόημα εάν θέλουμε πράγματι να καταπολεμήσουμε την, τις διακρίσεις βέβαια. ζητούμε λοιπόν αυτές τις τεχνικές πτυχές. Τις αναφέρατε και στα σχόλιά σας. Προθεσμία για τροπολογίε έχουμε τα τέλη Αυγούστου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Τέλη Αυγούστου, αρχά Σεπτεμβρίου και ευχαριστώ του πάντες για την κατανόηση. La euh, λέει η πρόεδρο. αφού είπε η Πρόεδρος αυτά που είχε να πει η πρόεδρο, είπε η συγκέντρωση αυτά που είχε να πει η πρόεδρο, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Κατάθεση τροπολογιών 27 Αυγούστου με ηλεκτρονική υπογραφή, εξέταση 18 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 17 Οκτωβρίου και έτσι κλείνει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για να πάμε στο 26 όπου συζητούμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την, ε, προς την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας ενέργεια σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας που συντάσσει ο κύριος Μπίτσικοφερ ως προς την νέα εθνομηχανή της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της Ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Με τις τροπολογίες πιστεύω θα μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα που παραμένουν ανεπίλητα. Δημιουργία λοιπόν νέων θέσεων εργασία και προτεραιότητες τη Επιτροπή μα, όπου λέμε ότι θα πρέπει να περνάει η νέα εκβιομηχάνηση από επενδύσεις πιο πολλές, πιο εστιασμένες, διαφοροποιημένες καθώς χρειάστηκε να αναπτυχθούν βεβαίως νέες τεχνολογίες, αλλά δεν μπορούμε και να λησμονούμε την παραδοσιακή μας βιομηχανική κληρονομιά, αεροναυπηγική, χάλιβα και αυτοκινητοβιομηχανία, όπως και πολλούς άλλους τομείς. Ε, μέσα λοιπόν τα οποία θα μας επιτρέψουν να, να να ξανακατακτήσουμε τις ε, παλαιές αγορές αλλά και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο επίπεδο θα σημαίνουν ε, την έρευνα για νέα μέσα παραγωγής, την προαγωγή ενός ε, της Ευρώπης ως κέντρου παραγωγής, την προαγωγή ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την ευρωκατάτηση των νέων. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων ε, παγκόσμια εμβέλεια, στου τομεί που έχει δύναμη η Ευρώπη και μπορούμε να προσαρμόσουμε και να προσαρμοστούμε καλύτερα στην νέα βιομηχανική πολιτική. Μια μόνο θηριδική προσέγγιση λοιπόν, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα, τις πληροφορίες που χρειάζονται, να ενημερώνονται για το πόσο χρήσιμο είναι να διατηρήσουν τις ε, δραστηριότητες του μηχανικές μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια και, ή και να επαναφέρουν στην Ευρώπη τέτοιου είδους επιχειρήσεις ένα συμβούλιο για τις επιχειρήσεις με 2,5 δισεκατομμύρια 2014-2020 και άλλο ένα πρόγραμμα που πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ωφέλιμο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, να ενθαρρύνουμε το ανταγωνιστικό και επιχειρησιακό πνεύμα, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τις μικρομεσαίες να τις βοηθήσουμε να δρουν και έξω από τα σύνορά τους, να διευκολύνουμε στην πρόσβαση στην αγορά, να Συμπληρώσω επίσης ότι υπάρχουν και άλλες νομοδοτήσεις στην έκθεση Μπουτικό, Φερίμ, Κόιντα και το καθεξής και εμείς θα προσπαθήσουμε τις υπολογίες μας να μην ξεφύγουμε από το δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων ώστε να διατυπωθεί σαφώς το μήνυμα της Επιτροπής μας, δηλαδή ισχυρή βιομηχανική παραγωγή που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω από τους συναδέλφους τις προτάσεις τους για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον εισηγητή και τις σκέψεις που εκφράστηκαν για τη σημασία της ε, ε, βιομηχανίας και την ανάγκη για αναζωογόνηση βιομηχανίας στην Ευρώπη, η οποία βεβαίω δημιουργεί θέσει εργασία που χρειαζόμαστε, δεν πρέπει αυτόν τον ρυθμονούμε, υπάρχουν καινοτόμοι τομεί και θα πρέπει να τους ε, αναζωογονήσουμε ενθαρρύνοντας το επιχειρησιακό πνεύμα, οι επενδύσεις στην κατάρτιση και την πρακτική εξάρτηση ασφαλώς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είτε για το πολιτισμικό πλαίσιο, είτε για τον προπολογισμό 2014 τα συζητούμε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η το ότι δεν δόθη συνέχεια στην νομοθετική πρωτοβουλία του συναδελφού Αλεχάνδρου για ένα πολύ καλό παράδειγμα και υπόδειγμα κοινωνικού διαλόγου για τις μικρομεσαίες θα πρέπει βεβαίω η μηχανία μας να στηρίζεται σε ηγετικέ μορφές αλλά και σε δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα αντίξω αποτελέσματα της λεγόμενης γραφειοκρατίας. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να ασωματωθεί σε μια τροπολογία θα ήταν έρευνα και ανάπτυξη να επικεντρωθεί, αλλά αυτό όχι αποκλειστικά μόνο στην, ε, στους νέους τομείς, γιατί αφορά όλους τους τομείς η έρευνα και η ανάπτυξη και χάρη σε αυτός μπορεί να και για την ανάπτυξη αυτή χρειάζεται να ενισχύσουμε τον, ε, τα σχετικά κονδύλια. Ε, διεθνείς εμπορικές συναλλαγές φυσικά και σχέσεις. Και εδώ θα έλεγα να προσέχουμε λίγο, γιατί όλοι τρέχουμε να κάνουμε ελεύθερες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να σώσουμε και να αναπτύξουμε ακόμα την βιομηχανική μας παραγωγή. Πρόσφατες πρωτοβουλίε Επιτροπής έχουν εκδηλωθεί. Θα πρέπει να τις... τις ε, πρωτοβουλίες αυτές σε άλλους τομείς. Ο Επίτροπος Ταλιάνη επίσης έχει επαναλημμένο σημειώσει ότι δεν έχει αρμοδιότητες ε, που είχε τον πρώτο καιρό Επίτροπος Νταβινιό. Έτσι λοιπόν την Επιτροπή του, στο τομέα του Χάλιβα και του Άνθρακα ίσως θα ήταν καλό να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να απτυχθεί μια κοινή βιομηχανική πολιτική που όπως η κοινή γεωργική πολιτική θα μπορούσε να έχει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και ένα ρόλο συντονιστικό, μια πραγματική δράση για την αναδιατύπωση τη ε, βιομηχανία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Άλλοι που θέλουν το λόγο. Όχι. Κομισιόν. κανεί, Όχι. Θέλω, θέλω. Σύντομα. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Δύο-τρία πράγματα να σχολιάσω. Οι προϋποθέσεις πλαίσιου καλύπτουν όλους τους κλάδους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους παραδοσιακότερους τομείς. Επίσης, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες για την πρόθεση των προσόντων ανακλάδο και η χαμένη ιδέα κοινή βιομηχανικής πολιτικής κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων τομέων της ε, κοινοτικής πολιτικής. Ξεκινήσαμε και προχωρούμε. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώ το λόγο στον εισηγητή. κάνω την παρατήρηση αυτή μετά την παρέμβαση σε κομισιόν και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι στη γνωμοδότησή μα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δικασία που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή με τον τίτλο Fitness Check, που θέτει τον εξή κίνδυνο να επανεξεταστεί η νομοθεσία σε μια σειρά τομέων, περιβάλλον και αλλού, και που θα έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα του, του της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει και κοινωνική διάσταση που πρέπει να μας ανησυχεί. Κύριε Σίγητα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την παρατήρηση που μας κάνατε, για το fitness check. Ευχαριστώ την Κομισιόν, τον κύριο Νταρντέν. Je Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα Είμαι βέβαιος ότι έχουμε κοινή παραγωγική δουλειά με παραγωγικά αποτελέσματα. Περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια των, ε, και τι τροπολογίες των συναδέλφων για να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε στην γνωμοδότηση αυτή και για να τη συμπληρώσουμε δίνοντας στην Επιτροπή τις θέσεις μας. Ευχαριστώ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Ιουλίου. 12 εξέταση των τροπολογιών και συμβαστούν 18 ψηφοφίζουμε στις 25 γιατί η ΙΤΡΕ θα ψηφίσει στις 26 Σεπτεμβρίου στις 17 Οκτωβρίου. Πρώτο τελευταίο σημείο στην σε διάταξη. Δίνω το λόγο για το, άρθρο, για το σημείο 22 στον συνάδελφο Τσάμπα Σογκό για να μας πει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για την δημογραφία που είναι αντικείμενο των τριών τριλόγων. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Köszönöm szépen, elnök asszony, a harmadik tárgyalás volt, Τρίτη διαπραγμάτευση ήταν για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τα δημογραφικά θέματα. Συζητήσαμε για την έννοια πληθυσμός, σύνηθις κατοικίες, σημεία 18 και 19, και το άρθρο, ενώ συζητήσαμε και το άρθρο 4. Το άρθρο 7 και 8 προ συζήτηση και έγκριση, ενώ δεχθήκαμε την παρέκκληση του άρθρου 8α και τη ρήτρα εποπτείας. Στον τρίτο τρίλογο πετύχαμε συμφωνία βάσει των προτάσεων της Προεδρίας ενώ λάβουμε υπόψη και τα σχόλια των γλωσσομαθών νομικών για τα άρθρα 5 και 3, 4 και 3, 5. Ενώ είδαμε και το 4 στην αιτιολογική σκέψη και το 1-4 στην αιτητογραφική σκέψη και το 14-8. Θα γίνει και μια ακόμα συνδιαλλαγή το Σεπτέμβριο, πριν έρθει το κείμενο στην Επιτροπή ξανά. Ευχαριστώ. Euh, bien, ε, bravo, monsieur. Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε εισηγητά. Εγώ θα πρότεινα απλά δύο λόγια. Ευτυχώς δεν έχουμε τρίλογο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της Κορεπέρ που ελπίζω να είναι να δώσει αποτελέσματα. Έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, την κατάργηση των, ε, ε, των ε, διαλόγων που περιλαμβάνει το, το Συμβούλιο και το ότι η διαβούλευση των νέων σημείων στον ερωτημάτων δεν θα γίνεται μόνο με διαβούλευση με τα κρατημέρια, αλλά θα εμπλεκόμαστε κι εμείς. Επί της ουσίας, να τονίσουμε ότι η δυναμική που θέλησε να παροτρύνει με το κείμενο αυτό η Επίτροπη που είναι να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα της κίνησης πληθυσμού λαμβάνεται παρκώς υπόψη παρότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Υπάρχει ιδέα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα παρακινεί τα κράτη-μέλη να μετράν καλύτερα τον πληθυσμό τους και για να λάβουν υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού στην στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο και για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι κάτι που με θλίβει ιδίω είναι ότι η λογική αυτή εφαρμόζεται τα δύο πεδία που ορίσαμε, δηλαδή το βάρος κάθε κράτους μέλους στο Συμβούλιο και την κατανομή των κοινοτικών πόρων, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αλλά ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται για τον καθορισμό του αριθμού των βουλευτών του κοινοβουλίου μας. Αυτό είναι συνεπές. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά μπορεί κάτι να χάσα. Θα, τα... θα επανέλθουμε το Σεπτέμβρη για να, για να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό μετά από εξέταση κορυφαία. Τελειώνουμε με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. 27. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και τους ευχαριστώ που ήρθαν. Δεν είχαμε δει μια συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων να κλείνει. Με χαρά σας καλωσορίζουμε Λίγο χρόνο μόνο μετά τη σύναψη της συμφωνίας που έγινε για το πλαίσιο, στο πλαίσιο της δράσης για την απασχόληση νέων και που αναφέρθηκε άλλωστε πριν από λίγο η Λιθουανική Προεδρία. Όσοι ήθιστε θα δώσω το λόγο τον Μαξίμ Σεργούτη, Business Europe κάναμε μία κατανομή του χρόνου εργασίας για να λάβουμε υπόψη το βάρος του καθενός, δηλαδή το πολιτικό βάρος, όχι το πραγματικό. Θα μας πείτε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συμφωνίας και τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να βοηθήσει τη δυναμική που προκύπτει. Κύριε Τσερούτη, 7 mm-hmm. λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Ε, θα παρουσιάσω τις ε, δράσεις για την απασχόληση των νέων. Οι διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο δράσεων ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2012 και καταφέραμε να τις ολοκληρώσουμε τον Απρίλιο του 2013. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι μέσα σε 7 μήνες ε, μπορέσαμε να πετύχουμε συμφωνία. Νομίζουμε ότι είναι μια ισορροπημένη συμφωνία, καλή συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική εταίροι συμβάλλουν στις λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Από πλευράς ε, των νέων ε, εντοπίσαμε διάφορες λύσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο. Χάρη στα μέλη μας και στο γεγονός ότι έχουμε μέλη από όλα τα κράτη αλλά και από τους οργοδότες και από τα συνδικάτα ε, διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο. Ε, προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω στις εφιστάμενες πρακτικές, να δημιουργήσουμε νέες, καλύτερες πρακτικές, ώστε και οι χώρες και οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται και τα Εθνικά Κοινοβούλια βεβαίως ε, και η Ευρώπη επίσης και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ άλλωστε. Πιστεύουμε ότι η εμβάθυνση όλων αυτών των πρακτικών θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε καινοτόμους τρόπους ε, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Από την πλευρά του Business Europe ε, θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο δράσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, η χρονική στιγμή στην οποία ε, συμβαίνει είναι σημαντική. Είναι μια πολύ καλή συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας, αλλά ανακοινώθηκε πρόσφατα στη Λιψία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγυήσεων στους νέους, εξίσου ε, πρόσφατο και σημαντικό. Ε, όλα αυτά έχουν, ε, θα έχουν μια συνεισφορά πολύ συγκεκριμένη και θα μας βοηθήσουν. Το πρωταρχικό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης νέων και αυτό είναι προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειάζονται ε, στεναρές μακροοικονομικές πολιτικές και βεβαίως αυτό μας απασχολεί. Ο ρόλος της ε, πολιτικής απασχόλησης και της ε, πολιτικής για την παιδεία είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τονίσαμε ε, την ανάγκη να έχουμε ανοιχτή και δυναμική αγορά εργασίας. Η σωστή εκπαιδευτική πολιτική και πολιτική απασχόληση θα συμβάλλει σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία θα βρήθει δουλειών που θα είναι πλούσια δηλαδή σε ευκαιρίες απασχόλησης. Η μάθηση ε, το χτίσιμο πάνω στις υφιστάμενες καλές πρακτικές. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Το πλαίσιο δράσεων έχει ένα κείμενο και ένα παράρτημα. Τα συμπεράσματα είναι στο παράρτημα. Π.χ. στη μαθητεία, το δανέζικο μοντέλο είναι μια πολύ θετική εμπειρία. Μεγάλο μέρος της μαθητείας λαμβάνει χώρα σε εταιρεία ε, στο πλαίσιο του μοντέλου διτής μάθησης. Ε, και θέλουμε αυτά τα συστήματα μαθητείας να εφαρμοστούν ενδεχομένως και σε άλλες χώρες. Ε, γιατί έτσι θα βοηθήσουν στο να βελτιωθούν οι ατέλειες του εκάστοτε συστήματος και αυτό είναι μεγάλο μέρος της απάντησης. Ασχολούμαστε και με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και μέσω της νομοθεσίας για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό, για να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νέους. Ασχολούμαστε ιδιαίτερως με το θέμα του εργασιακού κόστους. Καλούμε τους νέους να αναπτυχθούν μέσα στην αγορά εργασίας και κάτι που θέλω να τονίσω είναι μια σουηδική πρακτική, εξίσου σημαντική. Οι σουηδοί κοινωνικοί εταίροι στο τεχνικό τομέα και στο τομέα της μηχανικής γενικότερα, τεχνικοί και μηχανολόγοι Σουηδοί δηλαδή έχουν συμφωνήσει ε, για κάποιες λύσεις για τους νέους κάτω των 25 ετών. Όσοι λοιπόν είναι στη Σουηδία κάτω των 25 ετών και ενδιαφέρονται για αυτούς τους τομείς, οι Σουηδοί ε, κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να προβλέψουν μια ειδική σύμβαση εργασίας για αυτούς, διάρκειας 12 μηνών, η οποία μπορεί και να ανανεωθεί. Πληρώνεται ε, και δίδεται αμοιβή για την εργασία, για το χρόνο εργασίας, αλλά δεν πληρώνεται ε, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εισαγωγή σε μια εταιρεία. Ο χρόνος που περνάει δηλαδή ο εργαζόμενος μέχρι ότου να μάθει τη δουλειά και να μάθει τα της εταιρεία. Το εργασιακό κόστος είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό ε, και θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους και θα πρέπει να καταστήσουμε πιο ελκυστική την απασχολησιμότητα του νέου. Ε, τέλος, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό πνεύμα. Τονίζουμε το ρόλο της εκπαίδευσης για να καλλιεργήσουμε περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη και μάλιστα σε πρωταρχικά στάδια εκπαίδευσης και θέλουμε στοχευμένη στήριξη των νέων επιχειρηματιών. επιχειρηματιών. Έχουμε καλές πρακτικές π.χ. στην Ιταλία με το Talento Deleide, μια κοινή πρωτοβουλία της Κομφιτούστρια ε, των νέων ε, επιχειρηματιών και, της, ε, και μιας τράπεζας αυτή θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή πρακτική. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει διάφορες πρακτικές στο πλαίσιο δράσεών μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, ότι είμαστε συγκεκριμένοι, αλλά καλύπτουμε και το ευρύτερο ζήτημα της απασχόλησης ή της ανεργίας των νέων η μάθηση, η μετάβαση από τις σπουδέ στην αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό πνεύμα είναι τρία στοιχεία κλειδιά. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, αλλά θα πρέπει να λυθούν και τα διαρθρωτικά προβλήματα που κάνουν τη μακροχρόνια ανεργία των νέων στην Ευρώπη να παραμένει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Πρόεδρος, η διερμηνείς θα σας ευχαριστήσουν καθόλου γιατί ε, μιλήσατε εξαιρετικά γρήγορα, παρόλο που έτσι καταφέρατε να τηρήσετε το χρόνο που σας είχα δώσει. Πατρίκ από πλευράς ΕΤΟΚ, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Ευχαριστώ. Ο Μαξίμ το είπε. Δεν το είπε. Το πρόγραμμα εργασία ε, των κοινωνικών εταίρων που συζητήθηκε τον, Ιανου, τον Ιανουάριο του 2012 είχε εξ αρχής υπογραμμίσει μία υπερπροτεραιότητα Πρώτον, απασχόληση και ακόμη περισσότερο απασχόληση των νέων. Άρα έκανα τους υπολογισμούς στους 7 μήνες που διαπραγματευόμασταν, κάθε μέρα που πέρναγε, χίλιοι άνθρωποι, χίλιοι νέοι μπαίναν στους άνεργους. Χίλιοι περισσότεροι. Εξού και η πίεση. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις το φθινότερο του, του 12, αλλά στην πράξη επειδή υπήρχαν και άλλα θέματα για συζήτηση, η διαπραγμάτευση τους τρεις πρώτους μήνες ε, υπήρξε σημαντική εξέλιξη. Η συμφωνία πλαίσιο είναι η τρίτη τέτοια συμφωνία μετά το lifelong learning και την ισότητα. Εγώ θα έλεγα ότι οι συζητήσεις δεν ήταν εύκολες, ήταν πολύ ζωηρέ, πάρα πολύ μερικέ φορέ, αλλά συμφωνώ με τον Μαξίμ ότι είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση που μπορεί να τύχει υποστήριξη και εγκρίθηκε άλλωστε και από τα μέλη μας. Από πλευράς συνδικάτων είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 5 5.700.000 άνεργοι δεν μπορούν να ξεχαστούν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ελεγγύη μεταξύ των γενεών. Να αντλήσουμε από τους πιο έμπειρους, όχι τους πιο γέρους αναγκαστικά. Αλλά αυτό έχει επίπτωση στην κατανομή της ενεργείας. Μετά, όπως είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο, οι κοινωνικονομικές επιπτώσεις της κρίσης έφτασαν στα, τα όρια του κοινωνικά αποδεκτού σε πολλές χώρες. Ε, είναι γεγονός ότι πολλά μέτρα ήδη εγκρίθηκαν στον τομέα της απασχόλησης νέων. Η εγγύηση νέων για μας είναι ένα βασικό θέμα. Διότι συμβολικά οι τέσσερις μήνες οδηγούν σε εξελίξεις τώρα. Τα έξι δις, τα αρχικά 6 δις ήταν 166 ευρώ τον, για κάθε νέο, για κάθε χρόνο. Στη Γερμανία μόνο, για μαθητεία και μόνο, η, η χώρα δίνει γύρω στα 20.000 ευρώ τον νέο για να δείτε ότι τα έξι δις είναι ανεπαρκέστατα. Να μην μιλήσω για τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν για τη διάσωση των τραπεζών. Τέλος πάντων. Εμείς θεωρούμε ότι η προσέγγιση του κόσμου της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις, ναι, αλλά δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις προσδοκίες των νέων και να κάνουμε τους νέους σε τούβλα που θα πρέπει κάπως να τους ενσωματώσουμε για να ταιριάξουν σε αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις. Ναι, κινητικότητα, αλλά το να φεύγει σε ένα πληθυσμό 2.100.000 νέοι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί να λύνει ε, την, ε, το ζήτημα της ενεργείας, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ανάκαψη της χώρας συνολικά. Ποιότητα. Ποιότητα απασχόλησης, ε, μαθητείας, εκπαίδευση, σεβασμός των δικαιωμάτων βεβαίως. Παλέψαμε, αλλά τελικά βρέθηκε μια συνένεση, διότι κάποιες από αυτές τις θέσεις εργασίας, θέσεις μαθητείας μπορούν να αποτελέσουν ένα σκαλάκι για να προχωρήσουμε. Επιχειρηματικότητα. Ναι, επίσης, αλλά τονίσαμε ταυτόχρονα και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτά για τις προτεραιότητες από πλευράς μας. Είναι σαφές ότι σήμερα η κατάσταση είναι δραματική. Η σύναψη της συμφωνίας αυτής μέσω ενός σεμιναρίου είναι σημαντική. Τους επόμενους μήνες θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σε 12 χώρες φέτος και στις υπόλοιπες το 14 τη συμφωνία θα κινητοποιήσουμε τα μέλη μας για να δηλώσουμε μαζί, μας, μαζί σας τον πόλεμο, αν μου επιτρέπετε, να, να κηρύξουμε τον πόλεμο στην ανεργία των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Λιλιάν Μπολοζίνσκι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα και εγώ ε, να πάρω τη σκητάλη από τους δύο προλαλήσαντες. Η απασχόληση των νέων, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι κοινωνική, οικονομική αλλά και ανθρώπινη επίγουσα ανάγκη. Όλοι είμαστε περήφανοι γιατί οι διαπραγματεύσεις εξελίχθηκαν ταχύτατα. Μέσα σε επτά μήνες πετύχαμε πολλά σε μια πολύ καλή χρονική συγκυρία. Αντιμετωπίσαμε το θέμα της ανεργίας των νέων οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και μάλιστα δουλειά που να μπορούν να διατηρήσουν. Αλλά και οι εταιρείε δυσκολεύονται να βρουν νέους που να είναι κατάλληλοι. Έχουμε 80 συστάσεις, σωστά ισορροπημένες, με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τις απευθύνουμε στα κράτη-μέλη, στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, τους δημοσίους φορείς, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στις εθνικές αρχές τέσσερις προτεραιότητες. Εκπαίδευση, μάθηση, μετάβαση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις βασικές της τάσεις που για εμάς είναι υψηλής προτεραιότητας και για τους νέους αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως προς τη μάθηση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα προσοντούχων νέων Μάθηση που να έχει να κάνει με τη δουλειά, μαθητεία, στάζ. Ο Μαξίμ ανέφερε παραδείγματα. Σε χώρες όπου η μαθητεία είναι μακρά παράδοση, όπως είναι η Γερμανία ή η Αυστρία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπλέκονται ιδιαίτερως ως εκπαιδευτές, ως τρέινερ και χρειάζονται στήριξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προτείνουν νέες θέσεις ε, κατάρτισης εκπαίδευσης μαθητείας στους νέους. Green skills mismatches. Δεν έχουμε καλό τέριασμα μεταξύ ε, των δεξιοτήτων και αυτών που ζητάει η αγορά για να μπορέσει να υπάρξει μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία. Και θέλουμε εκεί να δουλέψουμε περισσότερο ώστε να καλύπτονται καλύτερα τα κενάνα και πρέπει να αναγνωριστούν περισσότερο και οι μη επίσημες δεξιότητες, τα μη επίσημα προσόντα. Αυτά θα είναι, αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τους ε, νέους με λιγότερα προσόντα. Είναι εξαιρετικά υψηλό το εργασιακό κόστος για τους νέους και υπάρχει και ακαμψία στην εργατική νομοθεσία πολύ συχνά. Ε, προτείνουμε συμφωνίες επί ειδικών όρων ώστε να έχουν οι νέοι πρόσβαση στην πρώτη τους δουλειά και να μπορέσουν να ενταχθούν με σταθερό, βιώσιμο τρόπο στην αγορά εργασίας. Και τέλος, επιχειρηματικό πνεύμα, κάτι το οποίο λείπει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι μια νοοτροπία που απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα, την επιχειρηματική κουλτούρα, ε, μέντορες να υπάρχουν ε, για τους νέους επιχειρηματίες. Ε, να έχουν αυτή τη στάση όχι μόνο οι νέοι που δραστηριοποιούνται ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, αλλά να έχουν επιχειρηματικό πνεύμα και οι εργαζόμενοι. Χρειαζόμαστε να είμαστε ευέλικτοι για να, να προσαρμοστούμε στις διαφορετικές εθνικές καταστάσεις, αλλά διαφορετικές καταστάσεις και σε επίπεδο περιφερειών. Όλες οι καλές πρακτικές πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους. Για να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο δράσεών μας θα πρέπει να υποστηριχθεί από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και από το σύστημα εγγυήσεων προς τους νέους, έτσι όπως έχουν αυτά ε, ανακοινωθεί από το Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι το σχέδιο δράσης για τους νέους της Επιτροπής θα εμπνευστεί από το δικό μας ε, πλαίσιο ε, δράσης και ε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και για να δεχθούν τους νέους. Τελευταία παρουσίαση. Ο Ανδρέας Πέρσον. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε το πλαίσιο δράσης μας. Στη συνέχεια του τι είπαν οι συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι τούτο αποτελεί μια σημαντική συμβολή των κοινωνικών εταίρων. Το πλαίσιο δράσεων περιλαμβάνει πολλούς τομείς μεγάλης σημασίας για τους κοινωνικούς εταίρους, τονίζοντας τομείς όπου χρειάζονται προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τρία θέματα θα σχολιάσω εδώ. Το σημαντικό θέμα της πρόθεσης της ελκυστικότητας και των σημαντικών εργασιών σε περιοχές έλλειψης, Φερρυπίν, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαψη, είναι θετικό. Ανά την Ευρώπη, πολύ... το δημόσιο τομέα συχνά σε πολλές περιπτώσεις ψάχνει κόσμο. Άρα η ελκυστικότητα των ε, θέσεων αυτών πρέπει να αυξηθούν. Αυτό ισχύει και για μελλοντικού τομεί όπου μπορεί να υπάρξει έλλειψη. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ εταίρων μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση και την ελκυστικότητα των θέσεων. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει το θέμα αυτό στο πλαίσιο δράση για την απασχόληση νέων. Η δυναμική εταιρική σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων μπορεί να γίνει με καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία, ε, εκπαιδευτικές δομές, σε open days για παράδειγμα. Επίσης η εμπλοκή των εταίρων μπορεί να βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές απασχόλησεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικής. Κάτι επίσης σημαντικό η επένδυση στην εκπαίδευση. Προφανές. Η απάντηση ωστόσο δείχνει ότι γίνονται περικοπές στην Ευρώπη. Η ανάγκη καλύτερης επένδυσης στην παιδεία είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Η οργάνωσή μου το καλωσορίζει. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση και τα συστήματα κατά της πρέπει να προχωρήσουν και να προσφυγούν για να δώσουν πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όσους τελειώνουν το σχολείο. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει αυτό το διαδικό σύστημα μαθητείας, παρότι πολλά χρόνια δείχνει πόσο καλή είναι αυτή η διαδικασία. Θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε προφανώς εσείς οι τέσσερις που εκπροσωπείτε τους ε, Ευρωπαίους συνομιλητές μας ως συντονιστής από πλευράς σοσιαλιστών ε, θέλω να σας συγχαρώ θερμά. Σταθήκατε στο ύψος των ε, ευθυνών σας σε μια τόσο δραματική στιγμή για την Ευρώπη και για το πιο ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού της. Πιστεύω ειλικρινά ότι το πρόβλημα δεν είναι των νέων, το πρόβλημα είναι δικό μας. Διότι, όπως είπατε και στην εξαρασία σας που κάνατε σε όλη την Ευρώπη, οι νέοι είναι το μέλλον μας και αν δεν έχουν μέλλον οι νέοι, τότε δεν έχει μέλλον και η Ευρώπη. Και από τη στιγμή που σε ορισμένες χώρες έχουμε ποσοστά αποτυχίας κατάφορης, έχουμε αποτύχει να ε, προσφέρουμε στους νέους ε, δυνατότητες να χτίσουν ένα μέλλον αξιοπρεπές, τελικά έχουμε οδηγηθεί στο να θυσιαστεί μια ολόκληρη γενιά. Και το γεγονός ότι μια ολόκληρη γενιά δεν θα μπορέσει να ζήσει θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, αλλά και δημογραφικά. Πώς μπορεί ένας νέος να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν ε, πάει στα 30, στα 35 και δεν έχει καν βρει δουλειά ή αν βρει ε, δουλειά έχει τόσο αβέβαιη ε, δουλειά και τόσο ε, καμιβόμενη... που δεν μπορεί να δεσμευτεί και να ξεκινήσει μια οικογένεια. Κανείς δεν το τολμάει. Είναι λοιπόν προβλήματα αυτά πολύ μεγάλα. Θέλω να σας συγχωρώ, να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας. Πιστεύω ότι η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο δείχνει ότι είναι μια ευκαιρία για τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν. Εμείς εγκρίναμε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να εργαστούν από κοινού με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, με τις επιχειρήσεις επίσης, για να υπάρξει κοινωνικός διάλογος. Οι χώρες που επιλύουν καλύτερα το πρόβλημα είναι οι χώρες ακριβώς όπου ε, είναι υψηλό το επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης και αναφέρομαι εδώ στην Αυστρία, στη Δανία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία και είναι υψηλό το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου. Σε αυτές τις χώρες λύνεται αυτό το πρόβλημα καλύτερα. Αυτές οι χώρες παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα. Η κοινωνία είναι σωστά διαρθρωμένη εκεί και οι νέοι δεν θεωρούνται ως ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, θεωρούνται ως ένα εργασιακό κεφάλαιο πάνω στο οποίο η χώρα πρέπει να επενδύσει. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιτυχία οι χώρες αυτές. Οι συστάσεις σα θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε όλους μας. Δεν έχουμε κάθε μέρα ευκαιρία ε, να ε, επιτυχάνουμε ε, τέτοιου είδους συμφωνίες κοινωνικές. Θέλω να ευχηθώ το καλύτερο για το Business Europe. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και να πω ότι μακάρι και στο μέλλον να πετύχουμε και άλλες συμφωνίες που θα μας διευκολύνουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μόνη αγορά, η μόνο οι επιχειρήσεις δεν αρκούν. Και πολλές περιπτώσεις μάλιστα χρειάζεται και συμμετοχή και ενεργητική συμβολή και άλλων ε, παραγόντων. Χαιρετίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες ως σοσιαλιστές, ωστόσο δεν επαρκούν. Αναφέρομαι στο σύστημα εγγυήσεων Εξαφανίστηκε βέβαια η λέξη Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησεων και δεν έχει και τους απαραίτητους πόρους η πρωτοβουλία αυτή ε, για να κάνει τη διαφορά στους νέους. Θέλω να εκφράσω και την ανησυχία μου ε, ως προς το εξής. Βεβαίως θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ή θέλουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες κατάρτισης. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν και είναι και πρέπει να είναι ένα πλαίσιο ποιότητας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μόνο μειώνοντας τους μισθούς, μειώνοντας τις παροχές, τις κοινωνικές, τις ασφαλιστικές κτλ. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα βραχυπρόθεσμα μόνο. Πρέπει να, ε, να έχουμε βάθος χρόνου, να κοιτάμε μακριά στον ορίζοντα και για να γίνει αυτό πρέπει να αποφύγουμε τις απλές και βραχυπρόθεσμες λύσεις και πρέπει να βάλουμε τη λέξη ποιότητα ε, στις δράσεις μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δεν μπόρεσα να διαβάσω το έγγραφο σε βάθος. Θα υπάρξει συστηματική συνέχεια, παρακολούθηση αυτού. Υπάρχει μηχανισμός ε, εποπτείας, παρακολούθησης. Γιατί αν ναι, μεταξύ ημών εδώ στο Κοινοβούλιο και ημών ε, μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό. Να το βλέπουμε, δηλαδή τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος και πώς ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πλαίσιο δράσεων οι διάφοροι ε, κοινωνικοί εταίροι. Δηλαδή, να δουλέψουμε όχι μόνο όταν ξεκινούμε τις πρωτοβουλίες και τις ανακοινώνουμε, αλλά και στη συνέχεια στη φάση υλοποίησής τους. Ε, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία ξανά να έχουμε διάλογο μαζί σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα. Υποσχέθηκα ότι θα μου λέω σίγουρα και στο συγγνώμη τους Ιρμηνές. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Πολύ ευπρόσδεκτο το έγγραφο. Εγώ ως Ιρλανδή έχω να επισημάνω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ιρλανδία και για την ενεργεία των νέων αλλά και με τη μετανάστευση όπου χάνουμε τους καλύτερους και πιο ικανούς νέους γιατί τους κερδίζει μετανάστευση. Και αυτό βέβαια όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγουν και το Καναδά, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για μας. Η ενέργεια αυτή έχει περαιτέρω αντίκτυπο και συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κυκλοφορούν άσκοπα στους δρόμους νέοι άνεργοι, γιατί αυτό βέβαια μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες. Όλα αυτά λοιπόν επιβαρύνουν πολύ την κατάσταση στην κοινωνία μας. Η προτεραιότητα που δίνει το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει και την προτεραιότητα της Ιρλανδικής Προεδρίας και με χαρά βλέπω μια συμφωνία 6 δισεκατομμυρίων για την ε, εμπροστοβαρή καταβολή της ε, εγγύησης για τους νέους. Όπως λένε όμως ότι άβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν. Και ρωτώ πώς ή σε ποιο βαθμό θα διαφέρει η εγγύηση για τους νέους από άλλα ε, μέτρα που έχουμε μέσα στο κοινωνικό ταμείο ή πώς μπορεί να στοχεύει κάθε κατηγορία αναγκών όταν αυτή τη στιγμή αποκλείονται από τα μέτρα του κοινωνικού ταμείου οι νέοι και όταν μπορέσουμε να τους πλησιάσουμε με το πρόγραμμα αυτό για τους νέους πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περάσει ένα εξάμεινο για να βρεθούν και πάλι στους δρόμους χωρίς καμία ε, διέξοδο και λύση όπου θα τους λένε παραδειγματί ότι δεν χρειάζονται πια. Θέλουμε η δουλειά να γίνει σωστά και να φέρει αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε ότι και από τις ε, όποιες καλές δουλειές έχουμε, οι νέοι μας τουλάχιστον στην Ιρλανδία, στο χώρο παραδείγματι των ε, νοσηλευτικών υπηρεσιών, ε, όταν βρίσκουν κάποια θέση εργασίας οι νέοι, είναι πολύ πιο χαμηλή αμοιβή η οποία τους προσφέρεται σε σχέση με, τα παλαιότερα, με το παλαιότερο προσωπικό και, δεν, και ως εκ τούτου αισθάνονται και εκτεθειμένοι απέναντι στα συνδικάτα τους, αισθάνονται δεν τους προστατεύουν τα συνδικάτα τους. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος που βρίσκει μία θέση εργασίας θα μπορεί να ε, τελειώνει μια κατάρτιση παραδείγματι, μια ε, πρακτική εξάσκηση και με μια πιστοποίηση που θα του επιτρέπει να βρει μια καλή θέση εργασίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν ε, να βρούμε λύσεις και σε ευρωπαϊκό, αλλά να κοιτάξουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε σε, σε εθνικό επίπεδο. Handel πρώτα και Ρέγκνερ μετά. Ναι, πολλά έχουν ήδη πει οι συνάδελφοι. Θα περιοριστώ μόνο σε, κάποιες βασικές, σε κάποια βασικά ζητήματα, το brain drain καταρχάς. Το περιέγραψαν οι συνάδελφοι, σημαίνει διαφυγή των ικανών νέων προς άλλες περιοχές, προς άλλους ε, προς άλλες χώρες του κόσμου. Και την ε, έλλειψη που γεννάται στις χώρες καταγωγής γιατί λείπει το δυναμικό αυτό, γιατί δεν καλύπτονται η ανάγκες από την παρουσία των νέων. Μια πρωτοβουλία λοιπόν για τους νέους ε, θα έπρεπε να σημαίνει και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. και να μην μείνει μεμονωμένη δράση. Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάξει πώς μπορεί με ολικά μέτρα να δώσει απάντηση στο πρόβλημα της ε, αλλά και της ε, ε, ανεργίας των νέων. Αυτό όλα τα λέω γιατί έχω υπόψη το πρόγραμμα αυτό, το πρόβλημα αυτό. Επίσης, βραχυπρόθεσμα μέτρα κατάρτισης θα μπορούσαμε να τα κοιτάξουμε με ένα κριτικό πνεύμα και να προσπαθήσουμε να τα ελέγξουμε και το λέω αυτό ε, συνειδητά. Διότι ασφαλώς ο κάθε εργοδότης θέλει φθηνό εργατικό δυναμικό και θα, θα πετάει τη σκούφια το άμα το βρει στη διάθεσή του. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν τα συνδικάτα σε όσες περιπτώσεις τι ρόλο παίζουν και όταν οι νέοι έχουν δυνατότητα κατάρτιση η οποία ε, έχει να τους προσφέρει όχι απαραίτητες ε, δεξιότητες, αλλά δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται ε, χρηστικές. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργούμε μία κατώτερη τάξη, συγχαίρομαι να χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, αλλά τελικά πρόκειται για μία κατώτερη τάξη, η οποία δεν έχει ελπίδα να ανέλθει οικονομικά και κοινωνικά. Επίσης στη Γερμανία ξέρετε ότι έχουμε μια μεγάλη παράδοση μέτρων τα οποία δεν αποτελούν ε, ουσιαστική κατάρτιση, μόνο στόχο έχουν να απασχολήσουν τους νέους, δηλαδή να μην τους αφήνουν στον δρόμο να κυκλοφορούν και δεν εξυπηρετούν τους στόχους πραγματικής κατάρτισης. Ας δούμε την πραγματικότητα στα μάτια. Αυτή η εγγύηση λοιπόν για τους νέους. Πολύ φοβούμε ότι εάν δεν μετατραπεί σε μια ουσιαστική πρακτική εξάσκηση και δυνατότητα επαγγελματική κατάρτιση, θα επιλέξει κατά πάσα πιθανότητα τον ίδιο ακριβώς δρόμο με το γερμανικό σύστημα, δηλαδή θα δίνονται κάποιες ε, το, θεσούλες ή κάποιες ε, δυνατότητες κατάρτισης μόνο και μόνο για να ικανοποιούνται οι στατιστικές ανάγκες χωρίς όμως ε, στοχευμένη αντιμετώπιση των αναγκών και των Χωρί μια άξια λόγου επαγγελματική κατάρτιση που θα επιτρέψει του νέους να βρουν μια θέση εργασία. Ευχαριστώ. Η επόμενη μου Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ίσως να είμαι η μόνη εδώ από την Επιτροπή μας η οποία τρέφει πραγματικές αμφιβολίες ως προς την εγγύηση νεολαίας. Εγώ ακούω τους νέους και ξέρω πολύ... Νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουμε το πρόγραμμα Εράσμους, το πρόγραμμα για τις δική των νέων. Νομίζω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε στο πρόγραμμα Εράσμου. λοιπόν. Είναι μια από τι μεγάλε επιτυχίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει ευκαιρίε στον νέο να αποκτήσει περισσότερε ευκαιρίε, περισσότερε εμπειρίε. Και πραγματικές πρόοδους, όχι οι πραγματικές δεξιότητες, όχι ε, αυτές ε, την ψευτοαπασχόληση που ανέφερε ο συνάδελφος νωρίτερα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε, και αυτή είναι και η ερώτησή μου, σε σχέση με τη δική σας εμπειρία, σε τι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα εγγύησης ε, νέων και όταν ε, δεν έχουμε τελικά τα αποτελέσματα τα οποία χρησιζόμαστε θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήσεις και μετά θα ξαναδώσω το λόγο. Ε, καταρχάς ε, για την μετανάστευση. Η ελεύθερη κυκλοφορία βεβαίως γράφεται στο επίκεντρο, είναι στον πυρήνα της συνθήκης της Ρώμης. Κανείς δεν αμφισβητεί την ελεύθερη διακίνηση, αλλά η συνθήκη της Ρώμης νομίζω ότι είχε υπόψη της μια κατεπιλογή ελεύθερη κυκλοφορία. Ενώ κάποιοι σήμερα μίλησαν για τον κίνδυνο της ε, ροής, έκροης ε, μυαλών. Ξέρουμε ότι στην Ισπανία παραδείγματι ένα ολόκληρο κίνημα αναπτύχθηκε και σύνθημά του έχει κάνει το «Δεν φεύγουμε εμείς, αυτοί μας διώχνουν». Εμείς στη Γαλλία στη δεκαετία του 70 είχαμε με επικεφαλής ε, το αριστερό συνδικάτο ένα ε, σύνθημα που ήταν να, να ζούμε και να δουλεύουμε στη χώρα μας. Πρέπει δηλαδή βεβαίως να υπάρχει κινητικότητα, αλλά άλλο κινητικότητα που έχει επιλέξει κανείς και άλλο κινητικότητα που, του, που την έχουν επιβάλει. Δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχρεώσει και να ορίσει κατά τρόπο δεσμευτικό τον τρόπο ζωής του καθενός. Όμως, ύστερα από τα όσα ακούσαμε από την συνάντηση, από το συνέδριο του Βερολίνου για την ενεργεία των νέων 3 Ιουλίου, θα πρέπει να διερωτηθούμε τι είδους μοντέλο μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί έχουμε αφενός και τη δημογραφική πίεση και την οικονομική πόλωση. Το καλύτερο μοντέλο ουσιαστικά θα ήταν οι νέοι πτυχιούχοι να ε, μπορούν να πάνε στις χώρες που έχουν πιο ηλικιωμένο πληθυσμό, πιο γυράσκοντο πληθυσμό, να βρούνε τις λύσεις που προσφέρονται και να δώσουν όσο μπορούν την ε, υποστήριξή τους. Όλα αυτά βέβαια που μπορεί να είναι detrimental θα έλεγα, δηλαδή μπορούν να αποβούν ε, εις βάρος των ε, νέων και εκπροσωπούν ένα κίνδυνο ουσιαστικά. Δεν έχω λοιπόν την εντύπωση, κοιτώντα το έγγραφό σας, ότι αυτή η διάσταση είναι παρούσα τόσο έντονα. Χρειάζονται ασφαλώς τα μέτρα τα οποία θα ασχοληθούν με τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες αλλά πέραν αυτού, η ανάπτυξη μόνη της δεν μπορεί να διορθώσει την πόλωση αυτή κατά τρόπο γενικό. Και επιπλέον ως προς την ε, συνέπεια της μετανάστευσης που επιφέρει για νέους, είτε ταλαντούχος είτε μη. Γιατί μιλάμε για δύο κατηγορίες νέων ουσιαστικά. Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο και τις συνέπειες του. Είπατε ότι έχετε κάνει μια καλή διαπραγμάτευση. Η ώρα εξέρχεται τρώγοντας όπως ξέρετε. Μας λέτε ότι επεξεργαστήκατε αυτήν την ε, συμφωνία. Υπάρχουν δυνατότητες και σε άλλους τομείς. Αλλά πέραν αυτού, ένας χρυσούς κανόν είναι το να κοιτάξουμε πώς αυτή η ποιότητα κοινωνικού διαλόγου θα φέρει αποτελέσματα εκτεταμένα, γιατί βλέπω ότι οι χώρες οι οποίες έχουν οικονομική ε, ευμάρεια είναι οι χώρες όπου ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί. Στις χώρες όμως που η Τρόικα έχει παρεύει δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος και προφανώς θα τον βελτιώνει και η Τρόικα με την παρουσία της. Πώς λοιπόν θα τα καταφέρουμε και λυπούμε που ε, διατυπώνω το ερώτημα αυτό σε τόσο προχωρημένη ώρα της συνεδρίασης, αλλά είναι ασφαλώς ένα στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί μιλούμε βέβαια για στόχους και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι μια πραγματική δυσκολία και παραπέμπει σε πρακτικές και συνήθειες και ιστορία, την ιστορία του συνδικαλισμού αλλά και της εργοδοσίας σε κάθε κράτος. Αλλά τώρα ξέρουμε πολύ καλά οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κατάρτιση, επαγγελματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, εγγύηση νέων κτλ. Όπου και να τα δείτε, σε όποια χώρα, αποτελέσματα φέρνει μόνο όταν υπάρχει κοινωνικός διάλογος. Εσείς λοιπόν τι μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό σαν ιδέα. Είπατε ότι θα κάνετε, ότι θα επισκεφτείτε τις πρωτεύουσε. Ίσως έχετε να προσφέρετε κάποιες ιδέες βέλτιστες πρακτικές. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να κοιτάξουμε και τη μεθοδολογία. Δεν βλέπω να ζητάει τώρα κανείς άλλος το λόγο. Ας ακούσουμε, όπως κάνουμε μερικές φορές, ανάποδα τώρα τους ομιλητές. Κύριος Πόρσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους βουλευτές που έκαναν σχόλια. Πολλές παρατηρήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντήσω για την ε, μετανάστευση και την διαρροή νέων ικανών. Χαίρομαι που αναφέρθηκε το θέμα αυτό, γιατί εμείς ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε αυτή την πτυχή ότι μετανάστευση ή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ε, πανάκια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα λύσει όποιο πρόβλημα έχουμε. Και αν κοιτάξετε, έχουμε διαφορούς τομείς, ε, όπως τον τομέα της ε, υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της Βαλτικής, όπου ε, φεύγουν πολλοί νέοι για να βρουν αλλού δουλειά και ως εκ τούτου βρίσκονται με σοβαρό έλλειμμα εργατικού δυναμικού σε νοσηλευτέ αυτοί οι τομεί. Για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, λοιπόν, ε, ναι, όταν υπάρχει ενεργεια 50-60% το βρίσκω φυσιολογικό να προσπαθεί κανείς ε, να βρει καλύτερες λύσεις. Και εμείς αυτές τις αρνητικές συνέπειες τις βλέπουμε συχνά και τις έχουμε υπογραμμίσει. Όσον αφορά την αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση της ε, ανεργίας των νέων, υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις, επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις, και επενδύσεις όπου μερικές φορές ε, δεν υλοποιούνται όπως πρέπει και οι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες των σοβαρών μέτρων λιτότητας στα διάφορα κρατημέλη. Ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου. Αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της ερώτησής σας. Ίσως θα μπορούσα να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια συστήματα όντως τα οποία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που παραμένει. Πολλές χώρες στο, στην περίπτωση του κοινωνικού διαλόγου έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις λόγω της κρίσης. Έκθεση παραδείγματι εργασιακών ε, σχέσεων ε, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία υπογραμμίζει τις διαφορές μεταξύ της ε, επιχείρησης να αντιμετωπιστεί η κρίση και των συνεπειών αυτής μαζί με κοινωνικούς εταίρους ή χωρίς. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχουν, υπάρχει κοινωνικός διάλογος το αποτέλεσμα είναι εποφελές ε, για κάθε πλευρά, για όλες τις πλευρές. Είναι λοιπόν ε, κάτι το οποίο σημειώνουμε και στις συλλογικέ συμβάσει και λέμε ότι μπορούμε ως κοινωνικοί εταίροι να προσφέρουμε πολλά. Αλλά δεν είμαστε εμονωμένοι παράγοντες. Πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να τοποθετηθούν και να συμπεριφερθούν ο λόγος στην υπόθεση αυτή. Αυτά και ευχαριστώ πολύ όλους όσοι έλαβαν το λόγο πιο πριν. Thank you, Madam Chair, being the second speaker. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στον κύριο Σέρκας για το πώς θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας. Στο πλαίσιο δράσης έχουμε μια διαδικασία ετήσιες εκθέσεως, αλλά θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. γι' αυτό ε, έχουμε κάνει σεμινάρια με συγκεκριμένους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνιτών τέρων για τον τρόπο υλοποίησης και για την βελτίωση των ε, δυνατοτήτων παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων. Μετά από τρία χρόνια ετησίων εκθέσεων θα κάνουμε και μία έκθεση αξιολόγηση. Δεν αφήνουμε λοιπόν τα μέλη μα ε, μόνα του, θα του βοηθήσουμε. Για τον τρόπο καλύτερης χρήσης της εγγύησης νέων. Αυτό που είπαμε είναι ότι χρειαζόμαστε να δώσουμε έμφαση στους νέους με τα σοβαρότερα προβλήματα. Την κατηγορία needs, ούτε απασχόληση, ούτε προσόντα δηλαδή. Στα αγγλικά είναι αυτό. Εκεί έχουμε και δυνατότητε με την εγγύηση των νέων και πολύ μεγάλη απογοήτευση και είναι οι πιο προβληματικές περιπτώσεις. Η δημιουργία μακροχρόνιας ανάπτυξη και εξέλιξη προς τις κρατικές αρχές θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη σοβαρά όταν θεσπίζουμε εθνικά προγράμματα δράσης χρησιμοποιώντας την εγγύηση νέων. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πλήρη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Χωρίς κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να έχουμε Ε, μέλλον ενδεχομένως να έχουμε και αντίθετα αποτελέσματα και μεγάλη απογοήτευση. Ο στόχος του, της εγγύησης νέων δεν πρέπει να είναι η βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφέρθηκαν ήδη τα προγράμματα Εράσμους, η κοινότητα των νέων, εμείς είμαστε υπέρ του Εράσμους Συν, του Erasmus Plus και την πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της κοινωνικότητας των νέων, αλλά όπως αναφέρθηκε, βλέπουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Είμαστε υπέρ των νέων για την ε, ε, απόκτηση εμπειρίας, αλλά και των νέων ε, και των νέων εργαζομένων. Όταν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και στον Νότο, την Ισπανία, ε, δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί που μετακινούνται φεύγουν. Α οι άνθρωποι κινούνται από μια χώρα σε μια άλλη, αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Δεν είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Ελπίζουμε ότι σε, με καλύτερες μακροοικονομικές συνθήκες και με καλή κατάρτιση. Δύο συνάδελφοι ήδη ανέλαβαν μας μια σειρά πρωτοβουλειών. Θα συνεχίσουμε στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε τη δύσκολη δουλειά. Τελευταίος. S'il me pas impossible. Euh, en ce qui concerne le suivi, Συνέχεια. Πρώτον, οι εσωτερικέ ε, σχέσει στο εσωτερικό τη ETUC και με τους εργοδότες το 11, έδειξαν ότι υπήρχε μία αίσθηση αποδυνάμωσης. Αν δείτε το πρόγραμμα εργασίας 2012-2013, πρόκειται για ένα από τα θέματα που αποφασίσαμε να δουλέψουμε. η οικονομική διακυβέρνηση η οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι παρά μόνο η πρώτη φάση. Μέχρι τώρα, μετά από την τέταρτη και τελευταία έκθεση, χανόταν το πλαίσιο δράση από τις οθόνες μας. Κανείς δεν το προσχεί και αυτό είναι επικίνδυνο γιατί όπως είπαμε και από πλευρά συνδικάτων δεν τίθεται θέμα να μετέχουμε στη δημιουργία μιας Ευρώπης τριών ταχυτήτων. Ευρώπη όπου οι συμφωνίες υλοποιούνται, συμφωνίες όπου δεν που δεν υλοποιούνται και χώρες που δεν γίνεται τίποτα. Εμείς έχουμε βλέπουμε ότι υπάρχουν συμφωνίες πλαίσιο που δεν υλοποιούνται σε, καμία, σε κάποιες χώρες. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς είπαμε ότι πέραν του τέταρτου έτους, σε χώρες που δημιουργούσαν προβλήματα, αν ήταν αναγκαίο, θα ξαναγυρίζαμε πίσω, θα με τους κοινωνικούς εταίρους, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, διότι έχουμε επίγνωση της προβληματικής στο capacity building. Πιστεύω ότι επιβεβαιώνουμε σαφώς μια σειρά συνθήκων, ε, άρθρων της συνθήκης και αυτονομίας των εταίρων. Δεν είναι δυνατόν η Τρόικα να έρχεται και να διαλύει με το α ή β πρόσχημα το κοινωνικό, το μας μοντέλο και τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι χώρες, και αυτό πρέπει να περάσει, ότι οι χώρες που αντιμετώπισαν καλύτερα την κρίση είναι οι χώρες που έχουν ισχυρή, ισχυρό πλαίσιο κοινωνικών, ε, κοινωνικού, διαλόγου κοινωνικών εταίρων. Βάσει των ετοιμάτων των κοινωνικών εταίρων ή όταν διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένους τομείς υπάρχουν ε, συγκρούσεις, προσπαθώντας να περάσουμε τις σωστές ιδέες με καλά αποτελέσματα μερικές φορές, διότι όταν ε, συζητούμε με τα προβλήματα αυτά σε πολλές χώρες, ε, επιτρέπουμε να ε, λύσουμε κάποιες παρανοήσεις. Το brain drain, τον, τον έφερε συνάδελφος, προφανώς δεν πρέπει να προσέχουμε γιατί ορολογία χρησιμοποιούμε. Ο Ανδρέας αναφέρθηκε στην κατάσταση σε μια χώρα της Βαλτικής, τότε υπήρχαν σαφή προβλήματα. Είχαν γίνει περικοπές στο δημόσιο, στην υγεία, με το υψηλότερο σήμερα ποσοστό θνησιμότητας, 42% παιδιών ζουν κάτω από το όριο φτώχειας, για την Τρόικα η κατάσταση ήταν καλή. Μείωσαν το έλλειμμα. Αλλά, so what? οι μεσοπρόθεσμες και σε επιπτώσεις ποιες είναι. Και σας το είπα ότι το συζητήσαμε με τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό, ξέρει ότι σήμερα μήπως θα έπρεπε, ξέρει ότι ε, μήπως έπρεπε σε, μια, σε κάποιες χώρες να σκεφτούν μια πολιτική ε, για τα συνδικάτα. Η δική μας αντιπροσωπή έχει νέους δώσαμε έμφαση στην ποιότητα της μάθησης. Βρίσκουμε τον όρο ποιότητα, προσφορά ποιότητας επίσης. Το Youth Guarantee είναι κάτι που το θεωρούμε σημαντικό. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να υπάρξει ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για, για την άσκηση. Ε, το, το Youth Guarantee δεν μπορεί να είναι ένα μια επιταγή εν λευκό για να κάνω ό,τι θέλουν οι επιχειρήσει Πρέπει να έχει όρους. Δεν είναι χρήματα για να απασχολείται ένας νέος έξι μήνες τελεία και παύλα. Αλλά και πάλι η κοινωνική εταίροι σε εθνικό επίπεδο θα συνεχίσουν τη συζήτηση που ξεκινήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επ' αυτού ακριβώς επειδή κυκλοφορούν διάφορες φήμες για ένα πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίξει τους ε, ασκουμένους ε, έχετε κάτι συγκεκριμένο, σκοπεύετε να επιληφθείτε ως κοινωνική Είπαμε ξεκάθαρα ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε. Είναι ιδιαίτερη διαπραγμάτευση γιατί είναι πολύ ειδικό το θέμα. Η πρόεδρος, άκουσα κάποιες φήμες ότι υπήρχε πρόβλημα από πλευρά κοινωνικών εταίρων. Δυσκολεύονται να προχωρήσουν στι διαπραγματεύσει. Επομένω, οι φήμε αυτέ ε, έχουν βάση. Νομίζω ότι εγώ πρέπει να απαντήσω, κυρία Πρόεδρε, λέει ο Μαξίμ. Εσείς το αποκαλείτε πρόβλημα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Για τη μαθητεία στο πλαίσιο δράσεων για την απασχόληση των νέων, ε, είχαμε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης, ασχοληθήκαμε με τη μαθητεία, με τα στάζ. Νομίζω ότι οι εργοδότες θεωρούν ξεκάθαρα ότι ε, στο πλαίσιο δράσεων πρέπει να ενταχθούν όλα αυτά τα θέματα. Εμείς έχουμε προβλέψει μια δυνατότητα να παρέμβουμε από κοινού μόλις υπάρξει πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα παρέμβουμε πριν παρουσιάσει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημειώνουμε, μας ενδιαφέρει. Απαντήσαμε ξεχωριστά γιατί τι είστε οι επόψει μας για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ε, νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα σχόλια. Θέλω να τονίσω κάτι που είπε και η κυρία Κοστέλο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και γι' αυτό οι συζητήσει είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι μπορεί να γίνει και θα έπρεπε να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Και θα σα δώσω δύο παραδείγματα. Η κυρία Βασιβέσκα ε, Μα είπε ότι έχει κάποιους, κάποιες αφιβολίες για την εγγύηση ε, προς τους νέους και η συζήτηση έχει εξελιχθεί εκ τότε. Υπάρχει μια σύγχυση ε, όρων Μιλούμε για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, η οποία ανακοινώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες από τον κοινοτικό προϋπολογισμό με συγκεκριμένο ποσό, το οποίο μάλιστα έχει αυξηθεί έκτοτε και ε, θα ε, μπει μαζί με νέους πόρους που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια απόφαση που λαμβάνεται σταδιακά, έχει σημειωθεί η πρόοδος και σιγά σιγά έχουμε φτάσει στα 14 δις με, την, ε, με το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, απαιτεί τη βούληση των κρατών μελών και έπαιξε και σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, η εγγύηση στους νέους είναι άλλο πράγμα, εκπορεύεται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ, και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τα κράτη-μέλη καλούνται να υιοθετήσουν μέτρα εξαιρετικά ευρεία μπορούν να είναι αυτά τα μέτρα για ε, δυνατότητες μαθητείας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ε, μιλούμε για προγράμματα ε, ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ε, απασχόληση νέων, ε, βοήθεια στους εργοδότες. Πολλά και διαφορετικά μέτρα εντάσσονται εκεί και οι συστάσεις δίνουν κάποιες ενδείξεις, κάποια παραδείγματα. τώρα, σε εθνικό επίπεδο για τις εγγυήσεις στους νέους, πρέπει να πω ότι η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από το ένα μέρος στο άλλο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η ανεργία των νέων είναι κάτω του 8% και η εγγύηση στους νέους δεν θα λάβει την ίδια μορφή με αυτή που θα λάβει στην Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων ε, είναι τεράστια και αποτελεί συστημικό κίνδυνο που υπονομεύει ε, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνία και την οικονομία, ούτως ή άλλως. Ε, προτείνουμε λύσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η συζήτηση για την εγγύηση των νέων είναι ένα παράδειγμα όλων αυτών. Στην εθνική συζήτηση για τις εγγυήσεις προς τους νέους θα πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα ότι τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συνεργαστούν για να ε, αντιμετωπίσουν τις βασικές προτεραιότητες που έχει το κάθε κράτος μέλος να τις ε, εφαρμόσουν. Άλλο παράδειγμα είναι το θέμα ε, της κινητικότητας και της διαρροής ε, εγκεφάλων, το brain drain, εν πάση περιπτώσει. Ε, είναι σημαντικό να πετύχουμε υψηλά επίπεδα κινητικότητας στην αγορά εργασίας κάτω του 3% των Ευρωπαίων κινούνται ε, υπό αυτή την έννοια, έχουν εργασιακή κινητικότητα, είναι κάτι που θα ευνοήσει την αγορά εργασίας, την οικονομία γενικότερα. Δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης δεν έχουν πληρωθεί σήμερα. Η αύξηση της κοινοτικότητας θα συμβάλλει στο να καλυφθούν αυτές οι θέσεις και να μειωθεί η ανεργία. Τώρα, άλλο είναι το θέμα του καταναγκασμού ε, ε, της ε, καταναγκαστικής κινητικότητας. Αυτό δεν αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όσοι φεύγουν από τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εκεί και αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συμφωνώ με την Λίλιαν δεν είναι μόνιμη αυτή η διαδικασία οι γλωσσικές δεξιότητες είναι επίσης σημαντικές. Βασική πρόκληση και εμπόδιο για την κινητικότητα είναι η γλωσσική εκπαίδευση αλλά και οι πολιτισμικές, οι πολιτιστικές διαφορές. Οι χώρες που στέλνουν εργασιακό δυναμικό στο εξωτερικό είναι αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αγορά εργασίας και πρέπει να δουν σοβαρά το θέμα, πώς θα μετριάσουν ε, τον αρνητικό αντίκτυπο των μαζικών αναχωρήσεων των νέων από την χώρα αυτή. Μπορεί να συζητηθεί και το, ο, ο κίνδυνος. Νομίζω ότι το εθνικό επίπεδο είναι το πιο κατάλληλο για να βρεθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στον κοινωνικό διάλογο και να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, για να είναι ο κοινωνικός διάλογος επικοδομητικός θα πρέπει να περάσει χρόνος. Ε, καλλιεργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Έχουμε κάποιες παραμέτρους ε, που συνδέονται περισσότερο με το θεσμικό πλαίσιο και βλέπουμε και πολλές διαφορές στην Ευρώπη σε ορισμένες χώρες επικρατεί η λογική του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και γι' αυτό και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν επιτυχία μεγάλη στον κοινωνικό διάλογο, δηλαδή και οι κυβερνήσεις σκανδιναβικές και τα κοινοβούλιο τα σκανδιναβικά θεωρούν ότι σε θέματα αγοράς εργασίας έχουν αρμοδιότητα πραγματική οι κοινωνικοί εταίροι και άρα έχουν και την ευθύνη να βρουν λύσεις, ενώ σε άλλες χώρους όπου οι δημόσιες αρχές έχουν αυξημένο ρόλο, ε, δεν το βλέπουν το πράγμα έτσι. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον κόσμο στον οποίο ζούμε είναι το εξής, ε, και στην Ευρώπη και αλλού. Ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι προσαρμόζονται στις ευκαιρίες. Είναι έτοιμοι να συζητήσουν τα πάντα το κόστος του συστήματος, τα θέματα ανταγωνιστικότητας των εταιριών, η ανάγκη ενίσχυσης ε, των δεξιοτήτων ώστε οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία κλειδί, ε, πολύ σημαντικά για την επιτυχία του κοινωνικού διαλόγου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τους τέσσερις ε, που ήρθατε μπορέσαμε να έχουμε μία άμεση ανταλλαγή απόψεων ε, για τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε κάπως ε, τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι υπέρ της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων Ως προς την οδηγία για το χρόνο εργασίας θα πρέπει να τονίσουμε την αυτονομία ε, των κοινωνικών εταίρων. Ε, με Βεβαίως αυτό ε, θα πρέπει να συζητηθεί και σε άλλη συνεδρίαση. Καλές διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.